Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινάμε. Ξέρω ότι εδώ και πολλά χρόνια είχαμε συνηθίσει να ξεκινάμε στις 3, τώρα ξεκινάμε μισή ώρα νωρίτερα και είναι δύσκολο να ξεσυνηθίσουμε, εξού και καθυστέρηση. Αλλά ας αρχίσουμε, να και είμαστε τώρα εδώ. Δεν είπα και τίποτα σημαντικό, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω αυτά που είπα πριν, ακόμη και αν δεν είχαν όλη τη ερμηνεία. Τώρα περνάω στα σημαντικά. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότατα στη συνεδρίασή μας τον κύριο Ρούμεν Ποροτζάνοφ, ε, Υπουργό Γεωργία Τροφίμων και Δασοκομεία στη Βουλγαρία, για μια ανταλλαγή απόψεων με θέμα τις προτεραιότητε τη Βουλγαρικής Προεδρία στο Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλώ ήρθατε κύριε Υπουργέ. Είχαμε συναντηθεί και με τους συντονιστές σήμερα νωρίς το πρωί. Και είχατε και πολλές ε, επαφές με μεμονωμένους ε, ευρωβουλευτές της Επιτροπής. Ε, είστε λοιπόν εκεί ο πρόσωπο για μας. Να σας υπενθυμίσω ότι το σύνθημα της Βουλγαρικής Προεδρίας είναι «Εν τη ισχύς» και αντικατοπτρίζει την ιδέα μιας Ευρώπης Ενωμένη αλληλέγγυα. Ε, κάτι που μας ενδιαφέρει και μας είναι και μα ιδιαίτερα προσφύλε θέμα. Θα μας παρουσιάσετε λοιπόν τις ε, προτεραιότητε και τα σχέδια της Βουλγαρικής Προεδρίας. Ε, θα μας πείτε τις απόψεις για την κοινή πολιτική μετά το 2020, το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, την ανακοίνωση του Επιτρόπου Χόγκαν της 29ης Νοεμβρίου αλλά και πολλά σημαντικά θέματα της αγοράς ε, με την κατάσταση να είναι σημαντική και ενδιαφέρουσα σε πολλούς τομείς. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη θέση των αγροτών στην τροφική αλυσίδα. Και υπάρχουν και άλλα επίκαιρα ζητήματα της γεωργίας που θα συζητήσουμε σήμερα. Πολύ σημαντικό θέμα είναι το πρόβλημα που απορρέει από την παγκοσμιοποίηση και τους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά λόγω της παγκοσμιοποίησης την ευρωπαϊκή γεωργία. Εσείς είστε η Δήμον όχι μόνο για τα θέματα της γεωργίας αλλά και για τα οικονομικά ζητήματα γιατί για πολλά χρόνια ε, ήσασταν σε πολλούς ε, φορείς και υπουργεία με τέτοιες αρμοδιότητες και σα ενδιαφέρουν και σας ε, αυτές οι διεθνείς συνθήκε και το πώς επηρεάζουν τα εσωτερικά μας. Επίσης σχέσεις ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Πάντω η γνώση και από οικονομικά θέματα και εμπορικά και η σχετική σα εμπειρία ενισχύει τη θέση σας ε, στη Γεωργία, γιατί γνωρίζετε πόσο σημαντικοί είναι οι εξωτερικοί παράγοντες. Σας συγχαίρουμε για την ανάληψη της Προεδρίας και σίγουρα εμείς θέλουμε να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε, να έχουμε αγαστή συνεργασία με την Βουλγαρική Προεδρία και μπορείτε να είστε βέβαιος ότι θα σταθούμε στο πλευρό σας. Ε, για σε αυτές τις τριγωνικές σχέσεις μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσπαθούμε να τονίζουμε την ε, ε, θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει νομοθετική αρμοδιότητα, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απρόθυμα μοιράζεται κάποια νομοθετικά προνόμια. Αλλά πιστεύω ότι η, συνεργασία μεταξύ μας θα είναι πολύ θετική. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα σε μια κρίσιμη στιγμή για την ανάπτυξη της ε, Γεωργίας και του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να σας παρουσιάσω τις ε, προτεραιότητες της πρώτης ε, Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το επόμενο εξάμεινο. Η Βουλγαρία θα είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι ένας καλός, καλόπιστος διαμεσολαβητής, συντονιστής και ηγέτης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συντονιστούμε, παρόλο που ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο. Ξέρουμε όμως ότι τι θέλουμε, ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε και ξέρουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ακούσουμε τις ανάγκες των πολιτών και να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις μετατρέποντάς τις σε ευκαιρίες. Στα πλαίσια της ε, τρέχουσας δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήθελα να, τονίσω την ε, σημασία της αγαστής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον ρόλο του ως συνομοθέτη και εκπροσώπου άνω των 500 εκατομμυρίων πολιτών. Και φυσικά θα ήθελα να εκφράσω την εγγνωμοσύνη μου για την υποστήριξη και που έχει λάβει και η ομάδα μου και εγώ προσωπικά από την ε, Επιτροπή σας στην προετοιμασία της σημερινής ακρόασης. Σας ευχαριστώ για την αρχική ανταλλαγή απόψεων που κάναμε και επίσης θα ήθελα να πω ότι είναι πραγματικά σημαντικέ οι προσπάθειε που κάνει η Επιτροπή σα ώστε να απλουστευτεί η κοινή αγροτική πολιτική αλλά και η ενεργό συμμετοχή σα είναι ιδιαίτερο σημαντική σε ευαίσθητου τομεί όπω η γεωργία, η, ε, ε, τα εισαγόμενα σιτηρά, η κτηνοτροφία κτλ. Ω πρόεδρο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλίας, εγώ από κοινού με τους άλλου θα προσπαθήσουμε να στείλουμε ένα ε, σημαντικό μήνυμα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τη, συμμετοχή, για τη σημασία συγγνώμη, της ε, ε, γεωργική πολιτική και της σημαντική προτιθέμενη αξία που έχει ώστε να παράσχει καλά προϊόντα στου πολίτες η Γεωργία μπορεί να συμβάλλει και στην αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή και φυσικά αυτό πρέπει να αναγνωριστεί από το κοινό. Και βεβαίω δεν θα πρέπει να υπάρχει αμφισημία μεταξύ τη ανάπτυξη γεωργία και τη διατήρησης του περιβάλλοντο. Επίση, η ε, συμμετοχή των νέων παραγωγών είναι πολύ σημαντική στην, στον τομέα τη γεωργίας και μάλιστα είναι και προπόθεση για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα και την οικονομία στι γεωργικέ περιοχές αλλά βεβαίως και τις οικογενειακές μικρές μονάδες στην ε, επαρχία. Πριν να αρχίσω να σας ε, παραθέτω τις προτεραιότητες μας για τους επόμενους έξι μήνες, να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου στην Εστονική Προεδρία για την πραγματικά εξαιρετική δουλειά που έκανε. Η Βουλγαρική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζεται ως μια ιστορική στιγμή, μεγάλη ευθύνη και μεγάλο προνόμιο θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις εταιρικές σχέσεις, τις συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, αλλά και αμοιβαία συνεργασία. Φυσικά θα προσπαθήσουμε με ε, επικοδομητικό τρόπο να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε απτά αποτελέσματα που θα έχουν όραμα προς το μέλλον, να διασφαλίσουμε την ε, λογοδοσία και την διαφάνεια και να είναι η Προεδρία μας ανοιχτή σε όλους τους πολίτες. Οι Ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται ασφάλεια και σταθερότητα και αλληλεγγύη, έτσι ώστε η ανταγωνιστικότητα, η ε, συνοχή είναι θέματα που θα απασχολήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο σταθερή και πιο ενωμένη. Επίσης θα προσπαθήσουμε να εξεύρουμε μια ισορροπία μεταξύ των συγκεκριμένων προτεραιοτήτων των κρατών μελών και, της, ε, και των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να έχουμε ε, ορατά και διαφανή αποτελέσματα στον διάλογο που κάνουμε με τους πολίτες. Και επίσης θέλουμε να απαντήσουμε και στις ε, ανάγκες που έχουν ε, οι πολίτες για βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, θέσεις εργασίας. Η Βουλγαρική Προεδρία θα προσπαθήσει να ε, δουλέψει πάνω στους τομείς της ασφάλειας, της νεολαίας, μέσα στο δεδομένο βεβαίως πλαίσιο που υπάρχει συγκεκριμένη προτεραιότητα της ε, Βουλγαρικής ε, Προεδρίας ε, έχει να κάνει και με τις προοπτικές των Δυτικών Βαλκανίων. Και επίσης η Βουλγαρία θα επικεντρωθεί και στην, ε, στις ευρωπαϊκές στρατηγικές προτεραιότητες, την, ε, την καλή γειτονία, τις καλές σχέσεις και την περιφερειακή συνεργασία. Είμαστε επιβεβαιωμένοι ότι οι ε, προτεραιότητες που έχουμε καταχωρήσει στο θεματολόγιό μας είναι σημαντικές και βεβαίως η εφαρμογή τους έχει να κάνει με την κοινή προσπάθεια όλων μας. Θέλουμε να επιτευχθούν οι στόχοι μας. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε επιλέξει το ε, ε, ενωμένοι ε, θα τα πάμε καλύτερα, είναι αυτό που πιστεύουμε βαθιά γιατί όντως αντικατοπτρίζει απολύτως μία ενωμένη και αλληλέγγυα Ευρώπη. Θέλουμε να δουλέψουμε λοιπόν ώστε να υπάρξει ενότητα μεταξύ και των ευρωπαϊκών κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων. Η Ευρώπη του αύριο είναι η Ευρώπη που θα αρχίσουμε να χτίζουμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε μια πιο ασφαλή ασφαλή και στέρη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα δείχνει αλληλεγγύη. Οι πολίτες περιμένουν να δώσουμε λύσεις στα προβλήματά τους. Η Βουλγαρική Προεδρία θα δουλέψει με διαφανή τρόπο και βεβαίως θα είναι ανοιχτή σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και σε όλους τους ευρωπαϊκούς εταίρους. Τρία βασικά είναι τα σύμβολα που αντικατοπτρίζουν ε, την, το λογότυπό μας, το οποίο προσπαθεί να δείξει ότι είμαστε ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης, αλλά επικεντρώνεται και στην μοναδική ταυτότητα που έχει η Βουλγαρία έναντι των υπολείπων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις κοινέ προτεραιότητες της ε, Βουλγαρικής Προεδρίας, θα ήθελα τώρα να περάσω στους συγκεκριμένους στόχους για την γεωργία. Ο εξυγχρονισμός και η απλούστευση της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής μετά το 2020 και ο προπολογισμό για τη γεωργία ε, με το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο είναι από τι βασικέ προτεραιότητε τη Βουλγαρική Προεδρία. Επί τη βάση τη ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον τη κοινή αγροτική πολιτική, θα οργανώσουμε μία σειρά συζητήσεων εντό του Συμβουλίου έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια καλύτερη κατανόηση των βασικών προβλημάτων και των στόχων που έχουν τα κράτη-μέλη. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ταυτόχρονα την ε, νομοθετική δουλειά. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να την καθοδηγήσουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και φυσικά αυτό θα συζητηθεί και στην ε, άτυπη υπουργική διάσκεψη στη Σόφια τον Ιούνιο του τρέχοντος. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διάφορες συζητήσεις που θα γίνουν, θα γίνουν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και κάποια τον Μάρτιο. Ο στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, σε κάποιους τομείς και να φτάσουν αυτά στο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δουλεύουμε πάνω σε πολλά θέματα κάποια έχουν συζητηθεί, κάποια όχι. Οι συζητήσει, ωστόσο, όπου έχουν γίνει είναι αρκετά γενικόλογε. Εμεί θέλουμε να επικεντρωθούμε στι άμεσε πληρωμέ, στη χρηματοδότηση. Θέλουμε να δούμε κατά πόσο είναι απαραίτητο να υπάρξει και έξτρα επιπλέον εθνική χρηματοδότηση που θα συμπληρώνει την ευρωπαϊκή, περιβάλλον, επικουρικότητα, και μάλιστα επικουρικότητα έτσι όπως ε, περιγράφεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ανακοίνωση αυτή μάλιστα μας δημιούργησε και κάποια ανησυχία σε σχέση με τις πιθανότητες που υπάρχουν για επανεθνικοποίηση των, ε, της ε, γεωργικής πολιτικής και γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Η πρώτη συζήτηση για αυτό το θέμα θα γίνει την επόμενη Δευτέρα. Επίσης θα μιλήσουμε για τα ανώτατα όρια για τις πληρωμές και επίσης ε, την μείωση των πληρωμών εφόσον έχουμε πετύχει κάποιο συγκεκριμένο κατόφλι. Ε, εκτός αυτού θα λάβουμε υπόψη και τις ειδικέ ανησυχίες και προβλήματα που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την χρονική διάρκεια όλων αυτών των συζητήσεων. Και επίσης θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τι γίνεται στις ε, γεωργικές αγορές, κυρίως για ευαίσθητους ε, κλάδους, γάλα, βοιοκρέας, χείριο, γαλακτοκομικά προϊόντα, φρούτα και λαχανικά και επίσης ζάχαρη μετά την απάλληψη των δασμών. Ε, επίσης θα δούμε και τις ε, ε, αθέμητες πρακτικές έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους παραγωγούς στην διατροφική αλυσίδα. Φυσικά περιμένουμε και τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας και θα προσπαθήσουμε να υπάρξει πρόοδος. Επίσης θα δούμε και τις ε, διμερείς και τις πολυμερείς συζητήσεις ε, και τον, ε, τους εμπορικούς διαλόγους και σε ό,τι αφορά τα δάση θα προετοιμάσουμε την πολιτική για την 13η Σύνοδο του, για το Φόρουμ για τα Δάση. Η Προεδρία θα δει ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι ώστε να προετοιμαστούν οι διαπραγματεύσει για μια δεσμευτική συμφωνία για τα δάση και επίσης θα προετοιμαστούμε και για την 24η Σύνοδο της Επιτροπής Δασών. Τώρα, για την ε, υγεία των ζώων, η Βουλγαρική Προεδρία θα επικεντρωθεί στην βιώσιμη διαχείριση της υγείας των ζώων και επίσης θα δώσουμε μεγάλη σημασία στην άγρια ζωή. θα επικεντρωθούμε στον αντίκτυπο, στις στρατηγικές για, την περιφερειακή συνεργασία, κοινή για άγριων ζώων. Θέλουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση της υγείας των ζώων σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Τον Μάρτιο του 2018 η Προεδρία θα οργανώσει ένα εργαστήριο για το ρόλο των αγρίων ζώων στην ε, υγεία των ζώων. Τώρα, για την ευζοία των ζώων, άλλη μια προτεραιότητα της ε, Προεδρίας μας, θα δούμε πώς μπορούμε να εναρμονίσουμε την τρέχουσα νομοθεσία. Επί τη βάση βεβαίως των όσων έχει κάνει η Εστονική Προεδρία, η δική μας Προεδρία θα δουλέψει μέσω τριμερών διαλόγων για τα γεωργικά στατιστικά, ελπίζοντας ότι θα έχουμε καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμβασμό που τελικά θα ικανοποιεί όλους. Σε ό,τι αφορά τώρα τα φυτογενομικά θέματα, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω στον σχεδιασμό των προγραμμάτων αντιμετώπισης και θα δούμε ποιε είναι οι δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκής Ένωση για τον έλεγχο και, την, ε, και τα φυτογενικά θέματα. Πρόεδρε, σας παρουσίασα κάποιου βασικούς άξονες της ε, Βουλγαρικής προεδρία και ευχαριστώ να απαντήσω και σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Πραγματικά ήταν ε, μεγάλη δόση πληροφόρησης που πήραμε. Θα θέλαμε λίγο χρόνο για να συνέλθουμε και να τα αναλογιστούμε. Αλλά αυτά, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να περάσουμε κατευθείαν στη συζήτηση. Πρώτος ζήτησε το λόγο ο κύριος Ντόρφαμ, που είναι ταυτόχρονα και εισηγητή ε, για την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Νοέμβριο, του 29 Νοεμβρίου. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας αξιότιμε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ για τα θέματα τα οποία θίξατε και τα οποία βεβαίως μας απασχολούν και μας στην Επιτροπή μας. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, μόνο κάποιες ε, ερωτήσεις για διευκρίνηση. Αναφερθήκατε στην ανακοίνωση του Επιτρόπου Χόγκαν και σε προσεχή συνεδρίαση του Συμβουλίου. Ε, μπορείτε να μας διευκρινίσετε παρακαλώ εν τέλει στο Συμβούλιο τι μορφή μπορεί να πάρουν τα συμπεράσματα, δηλαδή θα υπάρξει ε, τροποποίηση εκ μέρους του Συμβουλίου αυτού του εγγράφου, θα διατυπωθούν δηλαδή βάσει του εγγράφου αυτού προτάσεις του Συμβουλίου, βάσει της ανακοίνωσης, ή θα υπάρξουν και διαφορετικά θέματα, πέραν αυτών δηλαδή τα οποία αναφέρατε εσείς στα συμπεράσματα. Τοποθετηθήκατε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την επικουρικότητα. Όντως, ακούγεται πολύ ελκυστικός όρος ε, επικουρικότητα και βέβαια και στον τομέα των ε, ελέγχων έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η κατανομή λοιπόν αρμοδιοτήτων ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τοπικών ή περιφερειακών αρχών πρέπει να διαμορφωθεί κατά την άποψή σας διαφορετικά, πιο αποτελεσματικά, ώστε να ενισχυθεί και να απλουστευτεί βέβαια η επικουρικότητα. Γιατί φαίνεται αρκετά περίπλοκη αυτή τη στιγμή η εικόνα. Και εκεί όπου υπάρχει παρέμβαση στην αγορά, οι άμεσες ε, ενισχύσεις, δεν θα πρέπει να ε, αλλοιώνεται ο χαρακτήρα τη κοινή γεωργική πολιτική ω κοινή πολιτική. Να μην ξαναγυρνά δηλαδή σε εθνικοποίηση με την έννοια τη ε, παρέμβαση σε εθνικό επίπεδο του κάθε κράτους η γεωργική πολιτική. Μπορούμε να έχουμε μια ενιαία αγορά στα γεωργικά προϊόντα, στη γεωργική πολιτική συνολικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο δεδομένου ότι υπάρχει και ενιαία αγορά γενικότερα. Επίσης ε, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, όπως είπατε και εσείς, να ασκήσει πιέσεις ε, προς την Επιτροπή το Συμβούλιο ώστε στους προσεχείς μήνες να καταθέσει νομοθετική πρόταση. Ιδάλλως δεν θα προλάβουμε στην τρέχουσα θητεία του Κοινοβουλίου πριν τις ευρωεκλογέ να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και αποφάσεις για τα άγρια ζώα. Μιλήσατε για μια κατάσταση αρκετά δύσκολη αυτή τη στιγμή σε σχέση με, τον, με την πανόλη των χείρων, την αφρικανική πανόλη των χείρων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και εμάς. Έχουμε να κάνουμε και με φαινόμενα επιζωτιών που μεταδίδονται από το λύκο ή την αρκούδα. Πρέπει να τα δούμε λοιπόν. Επίσης μιλήσατε για φυτοπροστασία, ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, γιατί και χτες εδώ στην Επιτροπή μας είχαμε επιμακρών συζήτηση για το θέμα αυτό με πρόταση για νέους κανόνες και συστήματα αναγνώρισης και αδειοδότησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτό. Ο κύριος Ανδριού. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ που είστε εδώ στην Επιτροπή μας και εγώ έχω κάποιες σύντομες ερωτήσεις για να μπορέσουν όλοι οι συνάδελφοι να λάβουν το λόγο. Άλλωστε σας είδα και το πρωί. Πάντως ε, είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσει κανεί τον όρο κοινή γεωργική πολιτική αυτή τη στιγμή χωρί να αναφερθεί και στον προπολογισμό, μια και έχουμε τη συζήτηση εν εξελίξη για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, που όλοι γνωρίζουμε θα πρέπει μέχρι το Μάιο να οδηγήσει σε συγκεκριμένες αποφάσεις, όπως άλλως θεωρίζει το χρονοδιάγραμμα. Άρα λοιπόν, πριν μιλούμε για προπολογισμό για τη γεωργία, που θα θέλαμε βεβαίω να γνωρίζουμε και ποιε είναι οι θέσει τη ε, Προεδρία σα, ε, θα θέλαμε να ξέρουμε ποιε είναι οι θέσει σα συγκεκριμένα για την ε, προάσπιση του ευρωπαϊκού προπολογισμού στο πλαίσιο τη πολιτού δημοσιονομική του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Ποιες είναι οι δικές σας θέσεις λοιπόν. Είστε διατεθειμένος να συνοδεύσετε σε συγκεκριμένους όρους ε, και κονδύλια της προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ζητεί από το 1% να ανέβουμε στο 1,3% από ό,τι μας λένε οι πληροφορίες μας σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Αυτή είναι μια πρώτη ερώτηση που αποτελεί εκ των ονουκάνε φόρο ώστε να μην θυγούν και η κοινή γεωργική πολιτική και η πολιτική της συνοχής, οι δύο αυτές πολύ σημαντικές πολιτικές και βέβαια όλα τα ζητήματα τα οποία θίξατε στην ε, παρέμβαση σας. Έχετε κάποιες συγκεκριμένες και στεναρές θέσεις στην υπόθεση αυτή. Δεύτερον, στην επικουρικότητα και χωρίς να θέλω να επαναλάβω την ερώτηση του συναδέλφου Ντόρφμαν, θα σημειώσω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα. Έγινε λόγος για επανεθνικοποίηση, επαναφορά των αρμοδιότητων στα εθνικά κράτη-μέλη. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία στην επικουρικότητα ε, και σας ρωτώ συγκεκριμένα γιατί είπατε ότι χρειάζεται ένα σαφές πλαίσιο για την ε, ΚΑΠ στρατηγικό σχεδιασμό ε, αναφέρατε επίσης και περισσότερη επικουρικότητα ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για τα κράτη-μέλη. Ε, πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στο στάδιο στο οποίο έχουμε φτάσει πλέον. Δηλαδή στην ΚΑΠ θα αρκεί ε, να ορίζονται στόχοι μέχρι τις συγκεκριμένε δράσεις. Θα ορίζει η ΚΑΠ και τις δράσεις μας στα κράτη-μέλη ή θα περιοριστούμε στον προσδοσμό ή θα αφήσουμε στα κράτη-μέλη μεγαλύτερο περιθώριο ε, επιλογών και σε σχέση με τους στόχους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και από, αυτό θα, από την απάντησή θα εξαρτηθούν και οι μελλοντικές μας εργασίες βεβαίως. Ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θέλω καταρχάς να σας καλωσορίσω και να σας εκφράσω συγχαρητήρια και ευχές για την ανάληψη των καθηκόντων της Προεδρίας. Είναι ιστορική στιγμή για σας και τη χώρα σας ασφαλώς. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία λοιπόν στα καθήκοντα που έχετε αναλάβει. Στο εξάμεινο αυτό καθίσταστε και μέλος ε, της, ε, συμμετέχετε και στο δεύτερο σκέλος ε, των διαπραγματεύσεων για το Brexit. Εμείς, η περιοχή μου, η εκλογική περιφέρεια και η γενικότερη χώρα μου, έχουμε πια κουραστεί να ακούμε για Brexit και συνέπειες του Brexit, αλλά πρέπει οπωσδήποτε γιατί είναι ένα εξελίξει αυτή η διαδικασία. Οι συζητήσει που θα ακολουθήσουν στου επόμενου έξι μήνες ασφαλώς θα έχουν, ή 8 μήνες θα έχουν τεράστια σημασία για το μέλλον τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωση όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου. Εγώ προέρχομαι από την Βόρεια Ιρλανδία. Έχουμε αυτή τη στιγμή ε, σύνορα μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Δημοκρατίας Ιρλανδίας. Στις 30 όμως Μαρτίου του 2019 τα σύνορα αυτά είναι σύνορα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Το Δεκέμβριο το Συμβούλιο συνεδρίασε και πιστεύω πως όλες οι χώρες ε, δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να ε, παραγνωρίσουν τη σημασία του θέματος και να μπερδέψουν τις γραμμές. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα όσον αφορά τη γεωργία και την, ε, τις συναλλαγέ σε κυκλοφορία των γεωργικών προϊόντων από τι δύο πλευρές αυτών των συνόρων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη στις ε, συνομιλίες. Για τα όσα είπαν ε, οι κύριοι Ανδριού και Ντόρφμαν και το κομμάτι που αφορά τον προπολογισμό, εγώ είμαι ο αργιότερο εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας. Όταν ανέλαβα καθήκοντα ω βουλευτή, ε, η γεωργική πολιτική αντιστοιχούσε σε κομμάτι μεγαλύτερο από το 50% του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Τώρα έχει πέσει κάτω από το 40%. Και όσο προχωράει ο καιρό, Με ρωτούν βέβαια όλοι αν αντέχω γιατί συνεχίζεται αυτός ο αγώνας και η πίεση για μείωση της ε, αναλογίας από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό της γεωργικής πολιτικής. Είναι διαρκώς μειωτική η τάση. Ερωτώ λοιπόν πώς θα υπερασπιστείτε αυτά τα ποσοστά ε, και τον προπολογισμό για τη γεωργία με δεδομένα τα γενικότερα στοιχεία και τα πλαίσια μέσα στα οποία κινούμαστε. Και κάτι ακόμη. Υπάρχει ένας πυρετός επίτευξης παγκόσμιου εμπορικών συναλλαγών και εμπορίου και ειδικότερα αναφέρομαι στο Μερκοσούρ σας έχει κινήσει το ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση και κυρίως οι ανησυχίες κυρίως εκείνων που ασχολούνται με τα γεωργικά θέματα, ότι μια σειρά από εμπορικές συμφωνίες από την TTIP μέχρι κάθε άλλη ε, έχουν σοβαρές συνέπειες για τη γεωργία αλλά και τη βιομηχανία και φαίνεται ότι η γεωργία μετατρέπεται σε ε, αμνό προσφαγήν στην υπόθεση αυτών των συμφωνιών. Γιατί νομίζω δεν έχουμε περιθώριο να παραχωρήσουμε τίποτε άλλο σε αυτέ τι συμφωνίε. Δεν πρόκειται για Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται μετά για εμά που θα είμαστε εκτό με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να υπερασπιστούμε την κοινή γεωργική πολιτική και τα επιτεύγματα τη. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω τι απαντήσει σα. Ευχαριστώ κυρία Μιούλερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. ότι με Υπουργέ επιτρέψτε μου εκ μέρους της Γερμανίας να εκφράσω πρώτη τα... τις ευχαριστίες μου για τη Διεθνή Πράσινη Εβδομάδα. Είστε χώρα η οποία φιλοξενεί αυτή την εκδήλωση. Η Βουλγαρία έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση όπως και εσείς συγκεκριμένα σήμερα. Έχουμε να κάνουμε βέβαια με την κοινωνική πολιτική και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι από πλευράς Γερμανίας εμείς θεωρούμε ότι η επικουρικότητα για να είναι πραγματική θα σημάνει, για να υλοποιηθεί στην πράξη θα σημάνει ακόμη περισσότερη γραφειοκρατία ε, και πιο περίπλοκες ε, διαδικασίες από ότι ε, θα θέλαμε. Πολύ περισσότερο θα κινηθεί προς τις πιο περίπλοκες διαδικασίες και λιγότερο προς την απλούστευση. Πρέπει λοιπόν να δούμε συγκεκριμένα πώς μπορούμε στα επόμενα δύο-τρία χρόνια, πώς θα υλοποιηθούν οι προτάσεις, ώστε να είμαστε σε θέση να πούμε ότι πλέον έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Έχουμε ένα τομέα ο οποίο χρειάζεται ακόμη περισσότερη βελτίωση βεβαίω, αλλά πάνω απ' όλα δεν χρειάζεται να ανατραπούν τα πάντα στην κοινή γεωργική πολιτική. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια μετεξέλιξη, σε ήπιου τόνου. Και πιστεύω ότι αυτός ο πρώτος πυλώνας με τις άμεσες πληρωμές ε, θα πρέπει να αποβαίνει σε όφελος των μικρότερων επιχειρήσεων. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει και περισσότερη ή θα μπορούσε να υπάρξει περισσότερη αντικοποίηση και σε αυτό μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις γεωργικές. Θα το δεχθούμε και αυτό. Ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι αυτό, αυτό του διαλόγου με τους κτηνιάτρους και την κτηνιατρική και τα ζητήματα των επιζωτιών οι εμπορικές συμφωνίες και πάλι με το βλέμμα στη Μερκοσούρ μας γεννούν πολλές ανησυχίες. Ε, φοβούμαστε δηλαδή ότι θα θυσιαστεί στο βωμό της βιομηχανικής παραγωγής η γεωργία. Βεβαίως η Γερμανία έχει και σημαντικό βιομηχανικό κλάδο και ιδιαίτερα την αυτοκινητοβιομηχανία που θα συνεχίσει να πωλεί τα αυτοκίνητά της ανά τον κόσμο. Αλλά συγκεκριμένα εγώ θα ήθελα να γύρω το ζήτημα της μεταφοράς των ζώων και της ευημερίας των ζώων. Η Βουλγαρία, από ό,τι μαθαίνω, δεν έχει πολύ καλές επιδόσεις ως προς την ε, επιτήρηση των συνόρων της προς την Τουρκία στην υπόθεση αυτή. Πώς μπορούμε λοιπόν να ε, αποτρέψουμε τις, ε, σε μεγάλες αποστάσεις μεταφορές ζών των ζώων προς φαγή, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και βέβαια το θέμα της μεταφοράς του, των σφαγίων. Ευχαριστώ πολύ, Φλάναγκαν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και το θέμα του Brexit το συζητούν βέβαια σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά περισσότερο από οπουδήποτε άλλου, στην Ιρλανδία και βέβαια τη δημοκρατία σε σχέση με τις ε, συνέπειες που θα έχει για τη Βόρεια Ιρλανδία και τη δημοκρατία η επανεισαγωγή συνόρων, ε, όπως είπε και ο κύριος ε, Νίκολσον βεβαίως. Θα πρέπει πολλά πράγματα να τα κρίνουμε, να αποφασίσουμε και να επιλέξουμε για ορισμένα πράγματα στο εγγύς μέλλον. Και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω στο εξάμεινο που έχετε με αυτή την ισχυρή, με τη θέση ισχύω που κατέχετε αυτή τη στιγμή ως Προεδρία. Ε, θέλω να ρωτήσω λοιπόν το εξή γιατί με απασχολεί ε, δεδομένου ότι είναι αλληλοεξαρτώμενες η Ιρλανδία με το Ηνωμένο Βασίλειο και ιδιαίτερα στα θέματα της γεωργίας έχει πολύ μεγάλη σημασία η αμοιβαία εξάρτηση. Θα μεριμνήσετε εσείς ώστε η γραμμή των σύνορων να μην μετατραπεί σε γραμμή ε, κυρώσεων εις βάρος ε, των δύο αυτών ε, περιοχών της ε, Δημοκρατίας Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας με την εισαγωγή δασμών και ποσοστώσεων και μάλιστα σε μια περίοδο όπου ξεκινούν εμπορικοί πόλεμοι και εσείς είπατε ο ίδιος ότι δεν έφερε τα αναμενόμενα από πολλούς τουλάχιστον αποτελέσματα ο εμπορικός πόλεμος με τη Ρωσία. Μήπως λοιπόν, ε, μπορέσετε να, μήπως λοιπόν δεν μπορέσετε να κρατήσετε τις απαραίτητες αποστάσεις. Μήπως αυτό το κέικ το οποίο θέλετε να φτιάξετε ανακατευτεί με το λάθος τρόπο, γιατί βέβαια πρώτα πρέπει να ανακατέψει κανείς τα αυγά και μετά να προσθέσει το αλεύρι με τη σειρά. Μήπως λοιπόν η κουτάλα που κρατάτε μπερδέψει τα πράγματα. Μήπως πρέπει να έχετε υπόψη ότι αυτό το οποίο σκοπεύετε να βάλετε στο ταψί του φούρνου μπορεί να μας καταστρέψει με μια κακή συμφωνία δηλαδή για την Ιρλανδία και κακή συμφωνία και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχετε συνείδηση της σημασίας για μας αυτών των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ κύριε Σχόισλινγκ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε κύριε Υπουργέ να μας παρουσιάσετε το πρόγραμμα. Είστε σε μια καθοριστική σημασία ε, περίοδο ε, προεδρευών ε, καθώς ορίζονται τα ορόσημα για την κοινή πολιτική και το μέλλον της. Βεβαίω, ε, όπως είπαν και πολλοί άλλοι, τα πάντα θα κρυθούν από τα κονδύλια. Και βέβαια θα κρυθεί από το εάν θα μπορέσουν να διατεθούν τα κονδύλια εκεί που πρέπει, αν ο Γεωργός θα έχει την αίσθηση ότι παίρνει τα χρήματα τα οποία χρειάζεται όπως χρειάζεται, αλλά και ο καταναλωτής αλλά και το περιβάλλον, γιατί αν κοιτάξουμε τα ζητήματα του περιβάλλοντος, ε, το περιβάλλον, η βιοπικιλότητα, η όλη μας συμπεριφορά στη γεωργία μπορούν να επηρεάσουν πάρα πολύ το περιβάλλον, τις κλιματικές αλλαγές. Μίλησε ο κύριος Δόρφμαν για τα φυτοπροστατευτικά. Πρέπει δηλαδή να υπηρετήσουμε τους στόχους τους οποίους έχουμε ορίσει και με την τρέχουσα δημοσιονομική πολιτική. Αυτή είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε και νομίζω ότι η κοινή γεωρική πολιτική θα μπορούσε να κερδίσει και σε αξιοπιστία αν κάνουμε τι σωστέ επιλογέ. Πολλή λόγο γίνεται για τον πρώτο πυλώνα. Είναι πολύ σημαντικό όντω και καθοριστική σημασία ε, ζήτημα. Αλλά ταυτόχρονα είναι σημαντική εξίσου και η ανάπτυξη τη υπαίθρου. Δεν πρέπει να επιτραπεί δηλαδή περικοπή στο δεύτερο πυλώνα μεγαλύτερη από ότι θα βλέπαμε στον πρώτο πυλώνα και τι άμεσε πληρωμέ. Έτσι λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε όλο αυτό το εγχείρημα πριν από τις προσεχείς ευρωεκλογέ. και εδώ έχω πολλές αμφιβολίες διότι ο Επίτροπος είπε ότι το Μάιο θα καταθέσει προτάσεις ωστόσο ξέρουμε ότι χρειάστηκαν δύο χρόνια στις προηγούμενες ε, συζητήσεις για μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και τώρα μας λέει ότι μέσα σε 8 μήνες θα τα έχουμε καταφέρει. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Και πρέπει τα αποτελέσματα να είναι καλά ξεκάθαρα και να μας οδηγήσουν σε μια καλή μεταρρύθμιση. Ένα-δύο ζητήματα επίσης που θέλω να θίξω ε, που έχουν σχέση με τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Ξέρετε ότι η Επιτροπή μας ανησυχεί ιδιαίτερα και μεριμνά και για την ε, συμφωνία Μερκοσούρ. Ξέρουμε ότι συνεχίζονται στο περιθώριο και στους διαδρόμους οι συνομιλίες, το θέμα της Νέας Ζηλανδίας, Αυστραλίας, το βόλιο κρέας ε, και άλλα προϊόντα είναι επίσης πολύ επίκαιρα. Αλλά και το γάλα. Το συζητήσαμε ήδη ε, νωρίτερα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας κρίσης του γαλακτοπαραγωγικού τομέα. Ήδη οι τιμές στη Γερμανία καταπίπτουν, μειώνονται διαρκώς, ενώ έχουμε ακόμα περισσότερα ε, πλεονάσματα. Επομένως πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την προσεχή κρίση. Χρειάζεται κατεπηγόντως η απάντηση του Συμβουλίου. Η απάντηση αυτή η οποία θα μας επιτρέψει να αντιδράσουμε και να αντιδράσουμε εγκαίρως, όχι όπως πριν, με καθυστέρηση. Ευχαριστώ. Εσείς μιλήσατε για δύο. Κανονικά το μισό χρόνο δικαιούσασταν. Ο Άγνιο. Α, φαίνεται ότι δικαιούμαι 5 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα, όπως και προελήσατε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα τηρήσω, θα παίξω το παιχνίδι. Ε, είπατε, ο, είπατε κύριε Πρόεδρε ότι ο, ο Υπουργό τη Βουλγαρία ε, δεν ήταν μόνο Υπουργό Γεωργία αλλά και Δασοκομεία. Και έχουμε ένα πρόβλημα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί η δασοκομεία δεν εμπίπτει στι ε, κοινοτικέ αρμοδιότητε. Και η Επιτροπή τη Γεωργία ε, συντάσσει έκθεση πρωτοβουλία ζητώντα ε, ε, νομοθεσία για την δασοκομεία. Και πάμε στην Ολομέλεια και κάποια στιγμή θα έρθει και σε εσά το θέμα ε, κατά την Προεδρία σα. και φαντάζομαι οι 27-28 Υπουργοί Γεωργία θα αποφασίσουν ότι είναι εκτός θέματος αυτό το θέμα της δασοκομεία γιατί δεν υπάρχει κοινοτική αρμοδιότητα και θα λήξει και το θέμα. Αυτές οι βλακίες τώρα περί θέρμανσης του πλανήτη ή κλιματικών αλλαγών που σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσουν οι γεωργοί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ε, ε, ένα από το αέριο είναι το οξύδιο του αζότου και είναι υποπροϊόν της καλλιέργειας ψυχανθών. Ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ενισχύσει και να αυξήσει τις παρα... καλλιέργειες ψυχανθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αντίφαση αυτό. Ε, το έχω επισημάνει πολλέ φορέ και κανένα δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. σω θα χρειαστεί να το ψηφίσετε το επόμενο εξάμεινο. Επίσης αναφέρθηκε το θέμα της μικροβιακής αντοχής. Το είπαμε και στο πρόγευμα εργασίας που είχαμε το πρωί. Εγώ θα είμαι πιο θετικός. Ε, νομίζω ότι πρέπει να ανασκουμποθούμε γιατί αλλιώς θα χάσουμε πολλές ανθρώπινες ζωές. Και ελπίζω να... Εδώ πραγματικά είναι κοινό μας το πρόβλημα και δεν θα είμαι τόσο παρεμποδιστικός ο συνήθως ε, δεν θα κολλησιεργήσω. Τώρα για τις απαγορεύσεις των φυτοφαρμάκων, των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Πάντως κάποιοι υπουργοί γεωργίας ε, απήχαν ε, από τη στιγμή όμω που είναι Υπουργοί γεωργίας και ασχολούνται με τη γεωργία τη χώρα θα πρέπει να λάβουν μια θέση. Είναι υπέρ της απαγόρευση ή κατά. Δεν μπορούν να απέχουν και να σας φέρουν εσάς σε δύσκολη θέση ε, και να παραπέμψει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποχρεωθεί να έτσι να λάβουν απόφαση. Θα πρέπει επιτέλους να δείξετε πυγμή και να φέρετε πρώτον ευθυνών τους στους υπόλοιπους υπουργούς Υιοργών που δεν θέλουν να λάβουν θέση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Λαζό ε, όπως ξέρετε, οι χώρες Ανατολικής Ευρώπης ε, έλαβαν ενισχύσεις βάρος των χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Δεν είναι επίκριση αυτή, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων έδωσε 100 εκατομμύρια ευρώ δάνειο στην Βουλγαρία σε μια αγροφαρμακευτική βιομηχανία στα πλαίσια του σχεδίου Juncker. Και από το 2007 η προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ο τομέας των σιτηρών με τις ε, ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Η Ευρωπαϊκή ε, ένωση ουσιαστικά ε, αποδυνάμωσε τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπως ε, για το ΣΥΤΟ ενισχύθηκαν και βελτιώθηκαν οι υποδομές των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης με αποτέλεσμα να μας ανταγωνίζονται. 25% των σιτηρών παράγουμε. Έχουμε πολύ σημαντικό μερίδιο και επίσης ε, το μερίδιο της αγοράς που χάσαμε είναι αντιστρόφως ανάλογο από αυτό που κέρδισαν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτή είναι λοιπόν η συγκεκριμένη κατάσταση που ισχύει για τα σιτηρά σήμερα. Πρόσφατα ένας α, ε, α, ε, Γάλλος αγρότης εγκαταστάθηκε στην Ουκρανία γιατί θεωρεί ότι εκεί βρίσκεται το μέλλον. Εκεί είναι πολύ χαμηλότερο το κόστος και οι περιορισμοί πολύ μικρότεροι, πολύ λιγότεροι και είναι πολύ πιο ενδιαφέρον να επενδύει κανείς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί όμως έτσι έχουμε τον ανταγωνισμό. Και τον υποστηρίζει και έμεσα η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και έδωσε άδεια για την εισαγωγή Ουκρανικού ΣΥΤΟΥ. Πού είναι λοιπόν αυτή η αλληλεγγύη για την οποία μας μιλήσατε κύριε Υπουργέ. Επίσης μιλήσατε για απλούστευση της ΚΑΠ. Μακάρι να απλουστευτεί. Επίσης θα ήθελα να μου πείτε τι γνώμη έχετε για ένα σημαντικό θέμα, αυτό του αθέμητου ανταγωνισμού, αλλά και του χάσματο που δημιουργήθηκε μεταξύ της Χώρα τη Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να σταματήσει επιτέλους αυτή η σύγκρουση συμφερόντων που υπάρχει μεταξύ των χωρών τη Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριο Νέκοφ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Θα ήθελα και εγώ προσωπικά να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως θα ξέρετε, είμαι ο εισηγητής της Επιτροπής Γεωργίας ε, για τα διπλά ε, μέτρα και σταθμά στα προϊόντα της ενιαίας αγοράς ή τις ε, διπλές προδιαγραφές. Ποια είναι η γνώμη σας θα επιμείνετε στην συμπλήρωση της μεθοδολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την συνύπαρξη διαφορετικών προδιαγραφών μέχρι τα τέλη του 2018. Είστε υπέρ ε, ενός πανευρωπαϊκού φορέα που θα παρακολουθεί τέτοιου τους αθέμητες ε, εμπορικές πρακτικές όπως είναι τα διπλά πρότυπα. Επίσης, τα θέματα της ποιότητας των προϊόντων. Έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε ένα, μία από τις πρώτες χώρες που θα χρησιμοποιήσει τον όρο πολυπροϊόν. Μπορούμε να ε, υπολογίζουμε στη δική σας βοήθεια για να μπορέσουν οι παραγωγοί και σε ορεινές περιοχές που πραγματικά μοχθούν σε πολύ πιο αντίξωες συνθήκες γιατί το 40% των της αγροτικών, των αγροτικών εκτάσεων στη Βουλγαρία βρίσκονται σε ορεινές περιοχές να μπορέσουν να ορθοποδήσουν αυτοί οι άνθρωποι υπόσχεστε ότι μέχρι το ε, τέλο τη Προεδρία θα έχουμε καταλήξει σε μια πρόταση κανονισμού για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα ποιότητα, επίση είναι πολύ σημαντικά στι διαπραγματεύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τι λοιπέ χώρε, τρίτε χώρε. Και πολλά κονδύλια έχουν αφιερωθεί στην προώθηση των γεωγραφικών ενδείξεων. Και μάλιστα πριν από δύο χρόνια. Ε, Άρχισα να ασχολούμαι με τον εντοπισμό βουλγαρικών προϊόντων που ε, έχουν πιθανότητα να τύχουν προστασίας από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ποιότητας. Εσείς τι γνώμη έχετε, μπορούμε να εντοπίσουμε βουλγαρικά προϊόντα που να τύχουν τις προστασίες των γεωγραφικών ενδείξεων, μπορούμε να υπολογίζουμε στην ε, υποστήριξη στον τομέα αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα ποιότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις γεωγραφικές ενδείξεις και είναι και πολύ ε, ευαίσθητο στις διεθνείς διαπραγματεύσει που έχουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φάνταρ. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για την Εστονία. Είμαι εδώ εκπρόσωπος ε, των Εστονών ψηφοφόρων και χαιρόμαστε για αυτήν την αλλαγή της Κιτάλης από την Εστονία στη Βουλγαρία. Θα ήθελα να μας πείτε τη γνώμη σας για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, είστε ε, ε, επαϊόν και για οικονομικά ζητήματα, γιατί έχετε εργαστεί και στα Υπουργεία Εθνικό, Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας και γνωρίζετε το θέμα ε, της ε, διαχείρισης του κινδύνου στη χρησιμοποίηση των κονδύλιων. Ξέρετε πόσο σταθές είναι το κλίμα και όταν μια χώρα απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμπληρωματική ενίσχυση, εσείς τι γνώμη έχετε για τη σύσταση ενός ε, ενιαίου ταμείου διαχείρισης των κινδύνων, προκειμένου να επιληθούν τέτοιου είδους προβλήματα. Επίσης, ε, για την αλυσίδα εφοδιασμού έχω μια ερώτηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα των πληρωμών στα θέματα αυτά, αλλά το κύριο εισόδημα των αγροτών σχετίζεται με την αλυσίδα εφοδιασμού. Από εκεί αποκομίζουν το βασικό του εισόδημα. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε λοιπόν τη θέση του αγρότη, του παραγωγού στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ευχαριστώ κύριε δενανό, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ε, είμαι εισηγητής του θέματος ε, των φυτικών πρωτεϊνών και χαίρομαι που ε, θέσατε το ζήτημα αυτός προτεραιότητα της Βουλγαρικής Προεδρίας. Διεκπεραιώνουμε τώρα την έκθεσή μου που ευελπιστώ ότι την επόμενη εβδομάδα θα εγκριθεί στην Επιτροπή μας. Σίγουρα έχουμε τεράστια εξάρτηση για την εισαγωγή φυτικών πρωτεϊνών και σίγουρα η επισητιστική μας ασφάλεια και η βιωσιμότητα του συστήματό μας είναι το διοκύβημα αυτής της εξάρτησης. Χαίρομαι λοιπόν που ε, αναδείξετε ως προτεραιότητα αυτό το θέμα των φυτικών πρωτεϊνών και θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε και με τον όλο προβληματισμό για την κοινή γεωρική πολιτική. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια για να πείσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το θέσει ως προτεραιότητα της μελλοντική μας κοινή γεωρική πολιτικής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και οι υπόλοιποι παρακαλώ από ένα λεπτό καθένας. Ο κύριος Κουσμιούκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Πρόσφατα, στα τέλη του προηγούμενου έτους, ο Επίτροπος Χόγκαν, παρουσιάζοντας τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό, είπε ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές μια εξίσωση των αμέσων ενισχύσεων σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, εσείς ως εκπρόσωπος μια σχετικά νέα χώρας μέλους ε, ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα και ως υπουργό της Βουλγαρίας αλλά και ως Προεδρία. Οπότε φαντάζομαι η Προεδρία θα προετοιμάσει το Συμβούλιο για να λάβει παρόμοια θέση με αυτή που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εξίσωση των άμεσων ενισχύσεων σε όλες τις χώρες μέλη. Ε, φαντάζομαι ότι δύσκολο είναι να αποκτήσουμε τους υπόλοιπους. Αλλά οι ενδιαφερόμενοι πραγματικά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ο κύριος Βάιτς. Κύριε Υπουργέ, έχω διάφορα ερωτήματα να σας θέσω, πολύ σύντομα. Συγκεκριμένα για την επόμενη ΚΑΠ. Τα ανώτατα όρια ενίσχυσης ε, για τις βιομηχανίες θα τα προωθήσετε. Πρώτο ερώτημα αυτό. Δεύτερο ερώτημα, παρόμοιο με το συναδέλφο Μίλλερ μίλησε για τις, ε, τις μίλησε για, την, για τις μεταφορές ε, ζώων μεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας. Εσείς με τους ελέγχους των ε, μεταφορών τι θα κάνετε και με τη συχνότητα των ελέγχων, πώς πόσοι έλεγχοι θα γίνεται και πόσοι γίνονται ήδη. Και ένα τρίτο ερώτημα σε σχέση με την δασοκομεία αλλά και με την προστασία των περιοχών Natura 2000. Θα μπορούσατε να μας ε, παρουσιάσετε, να μας κάνετε μια δήλωση για το κατά πόσο αυτές οι κατηγορίες διαφθοράς σε ό,τι αφορά την, ε, την ε, διεύρυνση των περιοχών των πάρκων για σκι μπορούν να ξεκαθαριστούν. Και άλλο ένα ερώτημα σχετικό. Καταφέρατε την παράνομη υλοτόμηση σε τέτοιες προστατευόμενες περιοχές να τις σταματήσετε ή τουλάχιστον να τη μειώσετε. Και άλλο ένα σχόλιο, να σας ευχαριστήσω φυσικά για την ε, πολιτική που ε, ασκείται ε, απέναντι στην Μακεδονία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προς αυτό. Ευχαριστώ. κυρία ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ, κύριε Προεδρεύοντα και καλή επιτυχία στην Βουλγαρική Προεδρία. Κάποιοι προλαλήσαντες ε, κάλυψαν ένα τμήμα του θέματος, ε, γιατί πραγματικά στο εξάμεινό σας θα σας πέσουν δύο πολύ σημαντικά θέματα για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Καταρχήν, συζήτηση της ανακοίνωσης που μας έκανε ο Επίτροπος Χόγκαν και το θέμα της ρύθμισης ε, της τροφικής αλυσίδας. Γιατί το θέμα των τιμών παραγωγού είναι από τα μείζωνα θέματα και προβλήματα της γεωργίας. Χρειαζόμαστε μία ε, ευρωπαϊκή διάταξη και κανονισμό. Έχουμε εθνικές διατάξεις, αλλά δεν αρκούν. Χρειαζόμαστε μία ευρωπαϊκή κανονική, ε, κοινοτική ρυθμίση και υπάρχει σχετική δέσμευση. Επίσης θα πρέπει για όλα αυτά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα εριστικοποιηθεί να μην Ε, ακολουθήσει την κατάσταση των τεσσάρων από τις πέντε προτάσεις του Επιτροπού Γιατί συνήθως μιλούμε για δαπάνες μόνο της ΚΑΠ. Πότε δεν μιλάμε για έσοδα. Εγώ θα σας μιλήσω για τα έσοδα της κοινή γεωρικής πολιτικής και θέλω τη γνώμη σας. Εσείς ως μέλος ε, του Συμβουλίου και υπουργό ε, Εθνικός, τι γνώμη έχετε για τους ίδιους πόρους ή για την ενίσχυση της συμμετοχής ε, του Συμβουλίου στο επόμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί έχουμε νέες δεσμεύσεις, νέες πολιτικές. Πώς θα τις ε, εφαρμόσουμε με λιγότερα κονδύλια θα έχουμε και το χρηματοδοτικό κενό από το Brexit. Και να μας πληρώσουν τα διορθωτικά ταμεία και τα Ταμείο Συνοχής για να γεφυρώσουν το κενό δεν θεωρώ Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν νέα κονδύλια. Ποια είναι η γνώμη σας. Επίσης, το Συμβούλιο θα, θα λάβετε θέση επί της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και στην ανακοίνωση έχω, υπάρχουν δύο θέματα που με προβληματίζουν. Καλή επικουρικότητα, εκτός και αν με την ενοποίηση των πάντων ουσιαστικά επιδιώκεται επανεθνικοποίηση λόγω της συγχρηματοδότησης και σε αυτό διαφωνούμε. Έχουμε νέες προκλήσεις αλλά προσοχή. Θέλουμε μια κοινή γεωρική πολιτική. Και μέχρι στιγμής έχουμε μια πολιτική 28 χωρών. Εμείς ε, έχουμε, αν ε, έχουμε πανεθνικοποίηση, επειδή έχουμε αυτόνομες περιφέρειες, είχαμε 17 διαφορετικές προτάσεις για τη γεωρική πολιτική. Σε ό,τι αφορά τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Αναφερθήκατε και σε αυτό το θέμα και σας, ε, θα σας καλωσορίσουμε στον τριμερή διάλογο, αλλά θα πρέπει να γίνουν εκ παραλίλου οι συζητήσεις με το άλλο θέμα των κτηνιατρικών φαρμακοσκευάσματων, κτηνιατρικών φαρμάκων. Και τα δύο θέματα είναι αλληλένδετα. Έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε και να διεκπαιρεώσουμε τους δύο τριμερείς διαλόγους για τις φαρμακούχες δοτροφές και τα κτηνιατρικά φάρμακα. Τεκάστρο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, κύριε Προεδρεύον, για την παρουσία σας εδώ. Και ειλικρινά σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή επιτυχία στο εξαμεινό σας. Θέλω να επισημάνω τα εξή, ωστόσο, το ξέρουμε, θα το δούμε και στην έκθεση του αν θα γίνει και η παρουσίαση με την ε, κίνηση της συζήτηση σήμερα, ότι υπάρχουν ε, πολλές ανησυχίες ως προς την ιδέα αυτή για προτάσεις μεταρρύθμισης που θέλει να προωθήσει στους επόμενους μήνες ο Επίτροπος Χόγκαν. Πως μπορεί αυτή να αποκρύπτει ε, κίνδυνο επανεθνικοποίηση. Το είπαν πολλοί συνάδελφοι. Πού βρίσκεται λοιπόν η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ευελιξίας, επικουρικότητας για τα κράτη-μέλη, αλλά ταυτόχρονα ε, μη επανόδου στην επανεθνικοποίηση. Πρόκειται για μια ισορροπία που πρέπει να την ξανασκεφτείτε, να την ξανασκεφτεί το Συμβούλιο, που εμείς οπωσδήποτε θα ασχοληθούμε πάλι με αυτό. Ε, ταυτόχρονα όμως και το Omnibus και ξέρετε βεβαίως ότι έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια Κοινοβούλιο και Συμβούλιο για να συμβάλλουμε προς την απλούστευση με το, και το πρασίνισμα. Και δεν πρέπει αυτή η επικουρικότητα να μεταγραφεί σε περισσότερες περιπλοκές, σε πιο περιπλοκά συστήματα, και αυτό βέβαια μπορεί να προξενήσει τη μια μεγάλη, ιδιαίτερα σε χώρες που έχουν περιφερειακή οργάνωση, γιατί αυτό σημαίνει, ε, η επαναθνικοποίηση θα σημαίνει όχι ένα εθνικό σχέδιο, αλλά δεκάδες περιφερειακών σχεδίων που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ερωτώ λοιπόν που βρίσκεται αυτό το σημείο ισορροπία μεταξύ του κινδύνου τη επανεθνικοποίηση, αφενός και τη επικουρικότητας μαζί με την ευελιξία αφετέρου. Ευχαριστώ. Κύριε Σεράου Σάντο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, μα είπατε ότι δίνετε στο πρόγραμμά σας προτεραιότητα της, ε, τις αλλαγές ε, του κανονισμού Omnibus ε, στην ΚΑΠ και είπατε θα ασχοληθείτε με συγκεκριμένου τομεί. Αναφερθήκατε στο γαλακτοκομικό τομέα. Υπάρχουν ολόκληρε περιοχέ που εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από την παραγωγή γάλακτο. Όπω οι Αζόρε, για παράδειγμα, από τι οποίε κατάγομαι. Και είχαμε το κείμενο τη Άνοιξη ε, με αύξηση της παραγωγής ώστε να εξασφαλίσουμε την πραγματική βιωσιμότητα μετά την πρόσφατη διακύμαση των τιμών. Και μάλιστα έχουμε πολλές προσδοκίες ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίλυση του προβλήματος των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Ελπίζουμε το αποτέλεσμα να είναι αποτελεσματικό ώστε να έχουμε μια σωστή κατανομή των τιμών σε όλη την ε, αλυσίδα και μια δίκαια αμοιβή για τους γεωργούς. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για τα ενοπνευματόδη ποτά, τα αλκοολούχα ποτά, θα ήθελα να, να τονίσουμε ένα μήνυμα που έχει μεγάλη σημασία για την Πορτογαλία. Θα ήθελα να σταθμίσετε ε, τι ε, μοίρα θα έχει το ενόπνευμα του ζήθου, γιατί θα έχει η, η λύση που θα επιλέξουμε μεγάλη σημασία για το κλάδο. Και επίση, ε, σε ό,τι αφορά τον τρόπο γύρασης ε, των μπράντι, και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να, αυτά τα δύο σημεία να τα προσέξουμε στον κανονισμό για τα ενοπνευματότυπα. Ευχαριστώ. Κυρία Χόιμπουχ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Πολλέ ε, παρατηρήσει έγιναν και για την επανεθνικοποίηση και εμένα με ενισχύει ελαφρώ το θέμα αυτό η Κομισιόν και έχει κάποιους ε, δείκτες και στόχους, ε, τους οποίους όμως δεν είδα στο έγγραφο αυτό. Στην δική σας εκτίμηση δεν αναφέρεται τίποτα για το τι θα γίνει με τις χώρες οι οποίες δεν μπορούν ε, ή δεν θέλουν να επιτύχουν τους στόχους αυτούς ή δεν θέλουν να κάνουν τις κινήσεις προς την επίτευξη των στόχων αυτών. Υπάρχει κάποιος μηχανισμός κυρώσεων ή τι γίνεται με, τους, με τις χώρες αυτές. Θα ήθελα αν έχετε μια απάντηση παρακαλώ. Και επίσης το θέμα των αγορών θα ήθελα να υπογραμμίσω. Ο συνάδελφος Χόισλινγκ είπε ότι χρειαζόμαστε κάποια εργαλεία για την αντιμετώπιση κρίσεων. Μιλήσατε για τις συνθήκες και τις διάφορες συμφωνίες. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα αρκέσει ωστόσο. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε εργαλεία τα οποία να μπορούμε, με τα οποία να μπορούμε εκ των προτέρων να παρέμβουμε σε μια περίπτωση κρίσης. Δεν μπορούν να, να αναλαμβάνουν συνέχεια οι γεωργοί μας ή οι παραγωγοί μας να περνούν κάθε δύο ή τρία χρόνια τέτοιες ε, κρίσεις και να χάνουν και εισόδημα και παραγωγή. Ευχαριστώ. κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίαση του προγράμματος της Βουλγαρικής Προεδρίας για τη Γεωργία. Το, έχω ένα πρόβλημα με τα ανώτατα όρια των άμεσων ενισχύσεων. Ποια είναι η γνώμη σα ε, για το, αυτό το θέμα τη υπερξανότητα των ορίων για τι άμεσε ενισχύσει και τι γίνεται με την ε, γραμμικότητα των ε, ενισχύσεων, γιατί ο, η παραγωγή, οι αγρότες είναι σημαντική φορή τη ενιαία αγορά. Τι γίνεται με την ευθυγράμμιση λοιπόν ή την εξίσωση των άμεσων ενισχύσεων. Σε ό,τι αφορά τι σχέσει μα με τρίτες χώρες με μπλοκ χωρών όπως τη Μερκοσούρ. Υπάρχουν χώρες που επιθυμούν συμφωνίες εμπορικών συναλλαγών με τρίτες χώρες, αλλά όχι εις βάρος της γεωργίας. Δεν θέλουμε ποσοστώσεις κρέατος, βοήου για παράδειγμα, ή μοσχαρίσιο κρέατος από χώρες του, του Μερκοσούρ. Παρόλο που δεν είμαστε κατά το εμπόριο, γιατί είναι θέμα σεβασμού των προτύπων και προδιαγραφών ποιότητα. Θα ήταν αθέμητο ανταγωνισμό ει βάρο των Ευρωπαίων κτηνοτρόφων εισαγωγή τέτοιων προϊόντων και επίση θα διακύβευε την ε, υγεία των καταναλωτών στην Ευρώπη, όπω το κρέα από τη Βραζίλια που δεν θα τηρεί τέτοια πρότυπα. Κύριε κυρία Πετήρ, ευχαριστώ και θα ήθελα να σας καλωσορίσω κύριε Υπουργέ και να σας ε, ευχηθώ καλή τύχη στην Προεδρία σας. Τι γίνεται με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη RED 2. Εκεί έχουμε κάποιους κανόνες ε, για τη μελλοντική παραγωγή βιοκαυσίμων. Θα είναι προτεραιότητα της Βουλγαρικής Προεδρίας ε, ε, κατά το εξάμεινο αυτό, η οδηγία για τι ΑΠΕ, γιατί την περασμένη εβδομάδα το Κοινοβούλιο έλαβε θέση για το θέμα αυτό και ε, αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Επίσης μιλήσατε για πλούστευση της κοινή γεωργικής πολιτικής μετά το 2020 και αναφέρατε ως προτεραιότητα την ηλικιακή ανανέωση, την ανανέωση των γενναιών στη Γεωργία. Τι προτάσεις ε, θα υποβάλλετε για να στηρίξουμε τους νέους γεωργούς. Έχετε κατά νου κάποια μέτρα αποτελεσματικότερα από αυτά που είχαμε μέχρι στιγμής. Πρόκειται να προτείνετε κάποια μέτρα για τους πιο ηλικιωμένους γεωργούς ώστε να μεταβιβάζουν τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις σε νεότερους ε, όταν συνταξιοδοτούνται. Ευχαριστώ. Η κυρία Εράς Γκαρσία. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ στον ε, Υπουργό Γεωργίας της Βουλγαρίας ε, καλή τύχη Μακάρι να έχετε πολύ καλή τύχη στην Προεδρία σα. Έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτη αφορά την κοινή γεωργική πολιτική και την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύετε όντω ότι τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο θα δεχθούν ε, να στηρίξουν τόσο αμέριστα την ε, επικουρικότητα και επίση, πιστεύετε ότι μετά από 15 χρόνια που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μαλλιάσει να ζητάει ένα σχέδιο για την ενίσχυση των ε, ε, καλλιεργιών πρωτεϊνούχων ε, σπόρων. Θεωρείτε ότι εσεί στη διάρκεια της ε, Προεδρία σα θα καταφέρετε να υλοποιήσετε επιτέλου αυτή την υποστήριξη στην παραγωγή πρωτεϊνών. Σε ό,τι αφορά την τροφική αλυσίδα, ε, περιμένετε επιτέλους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πρόταση για την τροφική αλυσίδα, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ της κοινοτικής νομοθεσίας για τη ρύθμιση της τροφικής αλυσίδας, ώστε να αναχαιτιστούν οι καταχρηστικές ή αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Επίσης, το τελευταίο μου, τρίτο και τελευταίο ερώτημα αφορά τη σπατάλη των τροφίμων. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά μόνο στο πλαίσιο τη κυκλική οικονομία. Όλοι κοπτόμαστε, υποτίθεται, για τη σπατάλη των τροφίμων, αλλά την ώρα τη αλήθεια δεν κάνουμε και πολλά. Δεν είναι επαρκή τα μέτρα που έχουμε λάβει. Εσείς τι γνώμη έχετε και ως Προεδρία θα προτείνετε κάποιες δράσεις για να αποφευθεί η σπατάλη των τροφίμων στη διάρκεια του βουλγαρικού εξαμήνου. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Έχω μια ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Προέρχομαι από τις κατοχώρες και είδαμε εκεί ένα σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με μια απόφαση του Κοινοβουλίου που αφορούσε και την αλληλεία και επηρεάζει τις συζητήσεις που θα μπορούσαμε να έχουμε σε σχέση με τον Υπουργό Γεωργίας των Κατοχωρών. Εσεί, Εσείς λοιπόν αναλαμβάνετε ως περιοδικός προεδρεύων, δηλαδή για ένα εξάμεινο τα θέματα της Γεωργίας τα όσα είδαμε να εμφανίζονται τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες, τα fake news που τελικά οδηγούν ακόμα και τους βουλευτές να μην ξέρουν τι ψηφίζουν. Σας καλώ λοιπόν να συνεργαστείτε μαζί μας, να συζητούμε, να προετοιμαζόμαστε, να στηριζόμαστε σε δεδομένα πραγματικά και έτσι να και τι αποφάσει μα με τι ψηφοφορίε όπω έγινε και σήμερα. Διαφορετικά κινδυνεύει η ίδια η πολιτική γεωργία και ιδιαίτερα οι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει τη γεωργία. Θα ήθελα και εγώ να υποβάλω κάποια ερώτηση, κάποιες σκέψεις. Έχουμε επίγνωση της μεγάλη μεγάλης πολυμορφίας της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Α, συγγνώμη, ξέχασα τον κύριο Ροπέ. Προηγήστε κύριε Ροπέ. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė, iš tikrųjų išklausius jūsų. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα την παρουσίασή σας και τις προτεραιότητες σας και νομίζω ότι οι προτεραιότητες μας τελικώς είναι κοινέ. Το πιο σημαντικό τώρα είναι πώς θα καταλήξουμε σε συμφωνία για να τις εφαρμόσουμε. Όπως ξέρετε, το εισόδημα των γεωργών εξαρτάται από την τιμή και από την πληρωμή. Οι περιοχές όπου έχουν με χαμηλές τέτοιου είδους πληρωμές προφανώς έχουν και χαμηλές τιμές. Άρα δεν αξίζει να καλλιεργεί κανείς και έτσι οι γεωργοί μεταναστεύουν από τις περιοχές αυτές. Και μετά αναρωτιούνται εγώ πώς θα εφαρμόσω τα ευρωπαϊκά μέτρα με τόσο χαμηλές πληρωμές. Οι πληρωμές εδώ είναι πολύ χαμηλότερε από, ό,τι άλλες, από τις άλλες χώρες. Ε, νομίζω λοιπόν ότι αυτό το πρόβλημα πρέπει να το λύσουμε. Επίσης, το διεθνέ εμπόριο. Συνήθως η, ε, ενδιάμεση είναι αυτοί που ε, εκμεταλλεύονται και εποφελούνται τελικά και δεν νομίζω ότι ε, καταλήγουν τελικά τα κέρδη στους γεωργούς που ούτως ή άλλως είναι αυτοί που τα παράγουν. Και εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο συντομία. Γιατί είναι πολύ μορφή η Ευρωπαϊκή Γεωργία και αυτό είναι γεγονό. Υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία, υπάρχει διαφορετική γεωργία στο βορρά, στο νότο ε, και διαφορετικά επίπεδα προσλήψεων, διαφορετικά χαρακτηριστικά των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επίσης έχουμε νέε χώρε μέλη ε, με λιγότερο εξυγχρονισμένη γεωργία. Ε, ακόμη έχουμε κάποια κατάλοιπα της σοσιαλιστικής διάρθρωσης της γεωργίας και σταδιακά τα τροποποιούμε. Τι εργαλεία και μέσα μπορούμε να υιοθετήσουμε για να στηρίξουμε μια τόσο διαφοροποιημένη γεωργία. Δεν χρειάζεται να ε, εφαρμόσουμε μια μεγαλύτερη ελαστικότητα για να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στις χώρες. Ο κύριος Χόγκαν στην ανακοίνωσή του ε, λέει ότι η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση προσδιορίζει τους στόχους ε, και τις αξίες της κοινής διορικής πολιτικής και κάποιες, δίνει κάποιες οδηγίες, αλλά δεν υπησέρχεται στις λεπτομέρειες και τα κράτη-μέλη έχουν τη διακριτική ευχέρεια της υιοθέτηση των κατάλληλων μέτρων για την υλοποίηση των στόχων που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μάλιστα υιοθετούν και περιφερειακή προσέγγιση, γιατί ε, λαμβάνεται έτσι καλύτερη υπόψη ιδιαιτερότητα σε περιφερειακό επίπεδο. Οπότε υπάρχει ελπίδα στον τομέα αυτό με την ελαστικότητα. Επίσης, ε, το θέμα της γεωργίας ε, υποδεισμένης συνθήκες, ένδειξης συνθήκες. Αν δεν στηρίξουμε τέτοιες περιοχές, ορεινές, εξόχως απόκεντρες, θα ε, υποστούν μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση. Θα πρέπει να βρούμε ειδικού τρόπου στήριξη των ε, περιοχών με αντίξωε συνθήκε ε, για τη γεωργία, γιατί τέτοιε περιοχέ έχουμε σχεδόν σε όλε τι χώρε. Επίση, τι γίνεται με το γάλα ή με τι ζωοτροφέ. Γίνονται πολλές κερδοσκοπικές κινήσεις με τα προϊόντα αυτά. Θα πρέπει και αυτό να το αντιμετωπίσουμε Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί φορές που ασχολήθηκα με το θέμα αυτό. Τι γίνεται σε αυτά τα επίπεδα για αυτά τα εισοδήματα. Και τέλος, επιζωτίες ή επιβλαβείς οργανισμοί για τα φυτά. Έχουμε ασθένειες και στα ζώα και στα φυτά. Σε μεγάλο βαθμό είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις, αλλά δεν θα πρέπει να ενισχύσουμε την ετοιμότητά μας για να μην ερχόμαστε ε, εκ των υστέρων και να διορθώνουμε τα κακοσκήμενα πολύ αργά. Επίσης, είχαμε το πρόβλημα με τη Ρωσία, που είναι μεγάλος παραγωγός του υπουλερικών, χείριου κρέατος και κατάφερε να ενισχύσει και τη γαλακτοπαραγωγή. Και σε λίγο η ρωσική αγορά θα είναι κλειστή για τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα καμίας διείσδυσης των Ευρωπαίων παραγωγών στην ρωσική αγορά που όλο και κλείνει. Και οι κυρώσεις τελικά ε, δεν ήταν καθόλου αποτελεσματικές γιατί είχαν μόνο ένα πολιτικό χαρακτήρα. Ενώ οι Ρώσοι εφάρμοσαν εμπάργο που χτύπησε άμεσα τους Ευρωπαίους γεωργούς και χρειάστηκαν κονδύλια από τον κοινωτικό προπολογισμό για να σώσουμε την κατάσταση και να στηρίξουμε τους γεωργούς. Και Τώρα, αν είναι τόσο λίγο, δεν θα έχουμε πια δυνατότητα πρόσβαση στη ρωσική αγορά, γιατί δεν θα χρειάζεται τα ευρωπαϊκά προϊόντα η Ρωσία σε λίγο. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά. Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Бих искал благодаря за Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους για τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Η Βουλγαρική Προεδρία αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια δύσκολη περίπλοκη περίοδο και λόγω των εξελίξεων στην κοινωνική πολιτική. Και αυτό βέβαια θα απασχολήσει και τις μελλοντικέ προεδρίες, την Αυστριακή και τη Ρουμανική. γιατί και αυτές θα χρειαστεί να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά για να τα ε, ολοκληρώσουν, να ολοκληρώσουν τη μεταρρύθμιση. Άρα χρειάζεται να εργαστούμε πάνω σε μια πολύ σαφή γραμμή, με πολύ σαφές χρονοδιάγραμμα πάνω απ' όλα. Δεν μπορούμε να χάσουμε χρόνο. Πρέπει να οργανωθούν οι συζητήσεις ε, κατά τρόπο ικανοποιητικό Πρέπει να ξεκινήσουμε με δημόσιες διαβουλεύσεις βεβαίως, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής. Μετά πρέπει να συζητηθούν οι βασικές αρχές που περιγράφει η ανακοίνωση της Επιτροπής. Και Βεβαίως δεν υπάρχει θέμα επανεθνικοποίησης ή ανατροπής ε, των ισορροπιών ε, σε σχέση με την επικουρικότητα. Εδώ επιτρέψτε μου να διατυπώσω την προσωπική μου θέση. Ότι δηλαδή στους επόμενους 16 μήνες, στο διάστημα που μας μένει μέχρι τις ευρωεκλογέ, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και η νομοθεσία σχετική με την κοινή γεωργική πολιτική. Γιατί αν δεν έχει τελειώσει αυτή η δουλειά, και μέχρι τότε θα έχουν περάσει και δύο χρόνια που θα δουλεύουμε τα θέματα αυτά, θα είμαστε αναγκασμένοι να ξεκινήσουμε από το μηδέν, από την αφετηρία. Και ναι, διατέλεσα και υπουργό Οικονομικών. Γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν είναι καλό να επαναλαμβάνουμε τη δουλειά που κάνω ένας σε διαφορετικές θέσεις, να έχουμε επικάλυψη. Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που μεταλλάσσεται ταχύτητα, ταχύτατα, Υπάρχουν πολλές περιοχές ε, του κόσμου που δεν ακολουθούν τους δικούς μας κανόνες, που παραβιάζουν κάθε μορφής ε, διεθνούς, διεθνείς κανόνες, ακόμη και των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Αλλά αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει τη δική μας τη θέση για την νομοθεσία για το πολυμετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είπατε ότι όποιος ε, διαθέτει τα κονδύλια έχει και την εξουσία. Όντω συμβαίνει αυτό πάντα και παντού. Δεν είναι τυχαίο το ότι λέμε πως πρέπει να ενισχυθούν οι συνεισφορέ στον προπολογισμό δεδομένων και των ελλημάτων που αναμένεται να προξενήσει το Brexit αλλά και των αναγκών σε τομείς όπως η μετανάστευση και η ασφάλεια. καθώς θα χρειαστούν περισσότερα κονδύλια για τις πολιτικές αυτές δηλαδή. Οι πιο ογκώδεις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Συνοχή και η ΚΑΠ, αντιμετωπίζουν περικοπές. Και γι' αυτό προσδιορίσαμε και τη σχετική προτεραιότητα. Είχαμε και συνάντηση με τους υπουργούς πριν από μερικές ημέρες και προτείναμε αντιστοίχως ενίσχυση των ε, συνεισφορών των κρατών Όλοι οι συνάδελφοί μου λοιπόν, ακόμη και οι εκπρόσωποι των κρατηδίων της Γερμανίας, δηλώνουν πως πρέπει όντως να υπάρξει αύξηση των συνεισφορών προκειμένου να διαφυλαχθεί ένα κατάλληλο πρόσφορο επίπεδο χρηματοδότησης της ΚΑΠ και ότι ακόμη και αν υπάρξουν περικοπές, αυτές δεν πρέπει να έχουν σαν συνέπεια μείωση της ανταγωνιστικότητας για τα ευρωπαϊκά προϊόντα που κυκλοφορούν στις διεθνείς αγορές. Τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα είναι προϊόντα ύψης της ποιότητας που ε, την χάνουν πολύ υψηλή ζήτηση σε όλες τις αγορές του κόσμου και γι' αυτό έχει σημασία να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε βέβαια εμείς μόνοι μας να πάρουμε την απόφαση, αλλά εγείροντας το θέμα, ανοίγοντας τη συζήτηση στο Συμβούλιο των Υπουργών, εξηγώντας τη σημασία της διάστασης αυτής, πιστεύουμε και επιμένουμε ότι θα υπάρξει πρόοδος, πιστεύουμε και επιμένουμε οι συζητήσεις να γίνονται δημοσία, και κύριε εσείς, ο κύριος Ντόρφμαν ε, ρώτησε για, τις, ε, ε, για τα θέματα που μπορεί να συμπεριληφθούν κατά τις προβλέψεις μας τα συμπεράσματα. Ας δούμε τι θα προκύψει από τις συζητήσεις. Γιατί υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία συμφωνούν τα περισσότερα κράτη-μέλη, ενώ κάποια άλλα είναι πιο ευαίσθητα, όπως τα τα όρια, οι οροφές, η συνοχή κτλ. Βεβαίω τα νεότερα κρατημέλη μπορεί να θεωρούν ότι δεν είναι σε θέση να καλύψουν τα ποσοστά συγχρηματοδότησης όπως αυτά προβλέπονται. Εάν λοιπόν δεν αλλάξει αυτό, ποιοτική αλλαγή δηλαδή, δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα επιδοτήσεις στις άμεσες πληρωμές ή ενίσχυση εισοδήματος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να τα συζητούμε αυτά το ταχύτερο δυνατό και το αργότερα μέχρι το Μάρτιο να έχουμε ξεκινήσει ώστε να αποσταλεί και ένα σεφες μήνυμα προς τα θεσμικά όργανα το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή για το πόσο σημαντικό κρίνουμε το ζήτημα αυτό. Εάν μειωθεί στο μέλλον ο προπολογισμό για την κοινή γεωρική πολιτική, ε, αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο κατόπιν ενδελεχέστατης της ανάλυσης των συνεπειών για τον γεωργό, για τους διάφορους επιμέρους τομείς της γεωργίας. Γιατί υπάρχουν πολύ διαφορετικές συνθήκες αναλόγως του τομέα τη γεωργία. Δεν πρόκειται για το βόλιο κρέα, δεν πρόκειται για τα στηριά. Ε, οπωσδήποτε βέβαια, ό,τι και να κάνουμε, κάποιοι τομεί θα πληγούν. Και αυτό θα οδηγήσει σε οικονομικά αλλά και πολιτικά προβλήματα κάποια κράτη. Είναι δύσκολο να αποδεχθεί κανείς με τέτοια ανάλυση. Ωστόσο πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Πιστεύουμε ότι το πλαίσιο των συνομιλιών πρέπει να είναι ο προπολογισμό τη ΚΑΠ και για να περάσω σε κάποια άλλα ε, λεπτά ζητήματα όπως ε, τα, οι οροφές, το κάπινγκ, η ανακοίνωση της Επιτροπής ακροθυγώς μόνο αναφέρεται στο θέμα αυτό, δεν υπησέρχεται σε λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι κάποια κράτη-μέλη δεν επιθυμούν ε, τον προσδιορισμό των ορίων γιατί υπάρχουν ε, μεγάλοι συνεταιρισμοί εκεί με πολλούς γεωργούς, ε, όπου εάν πρόκειται για κάπινγκ ε, με το σύστημα του ενός αποδέκτη δικαιούχου, δεν μπορούν να έχουν ικανοποιητική χρηματοδότηση. Εμείς στη Βουλγαρία κάναμε την επιλογή του κάπινγκ με, την, ε, με τον προσδιορισμό μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ μεγάλων και μικρών παραγωγών και προχωρήσαμε και σε αναδιανομή των ε, πληρωμών. Βέβαια η συζήτηση είναι εν εξελίξη για το αν θα είναι υποχρεωτικό το κάπινγκ ή αν θα μπορεί το κάθε κράτος μέλος να λαμβάνει ε, τις δικές του αποφάσεις. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί από το μέλλον. Πάντως, είμαστε υποχρεωμένοι να ανοίξουμε το διάλογο αυτό, θα το πράξουμε. Εμείς προσωπικώς στους τρεις πρώτους μήνες της Προεδρίας μας σκοπεύουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση γιατί θέλουμε να είμαστε σε θέση ξεκάθαρα να δηλώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχουμε κάνει αυτές και αυτές τις επιλογές και εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ε, την επεξεργασία του θέματος πρέπει να γνωρίζει ε, μέχρι που είναι το Συμβούλιο να κινηθεί. Η Επιτροπή σας, ε, ξέρω ότι επεξεργάζεται μια έκθεση στο θέμα αυτό, που θα προωθηθεί για την ψηφοφορία στην Ολομέλεια το Μάιο, ε, μια έκθεση η οποία θα συμβάλλει και στην καταγραφή των διαφορετικών θέσεων και είναι πολύ σημαντικό να ετοιμαστεί πριν από την ε, κατάθεση των τελικών νομοθετικών προτάσεων. Και τώρα επιτρέψτε μου να περάσω σε ένα θέμα που ασφαλώς είναι πολύ ευαίσθητο. Το αναφέρατε ήδη. Επικουρικότητα και επανεθνικοποίηση. Εγώ προσωπικώς πιστεύω ότι δεν πρόκειται να γίνει η επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ, έχοντας μιλήσει μάλιστα και με εκπροσώπους κρατών μελών, διαφορών κρατών μελών. Θα επιμείνουμε βεβαίως να υπάρχουν σαφείς κανόνες και ένα κοινό πλαίσιο. Έτσι μιλούμε για μια κοινή γεωργική πολιτική. Και έτσι θα μπορούμε να μιλάμε για μια κοινή γεωργική πολιτική. Με το κοινό αυτό πλαίσιο θα έχουμε τη δυνατότητα της χρηματοδότησης κάποιων τομέων με κοινού και αυστηρούς κανόνες, οι οποίοι ωστόσο θα εφαρμόζονται με τρόπο λιγότερο δίσκαμπτο και άρα λιγότερο γραφειοκρατικό χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα είναι τέτοια η χαλάρωση των ε, ε, κανόνων που δεν θα ακολουθούνται αυστηρά κριτήρια για την διάθεση των κονδύλιων. Απλώς θέλω να επισημάνω ότι θα υπάρχει απλοποίηση μέσω των, θα προκύψει απλοποίηση μέσω των νομοθετικών προτάσεων. Και βεβαίως πρέπει να συζητηθεί η επικουρικότητα και η εντό εισαγωγικών επανεθνικοποίηση. Θα καταθέσουμε προτάσεις στο Συμβούλιο την προσεχή Δευτέρα. Αλλά υπάρχει κι άλλος ένας τομέας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός. Και πάλι για να αναφερθώ στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το στρατηγικό σχέδιο δηλαδή μπορεί να εξασφαλίζει μια δυνατότητα για επανεθνικοποίηση. Γιατί αφήνει πολλά ζητήματα αναπάντητα ζητήματα στα οποία εμείς πρέπει να δώσουμε απαντήσεις το ταχύτερο δυνατό. Ξέρω ότι έχουν ήδη συζητηθεί στην, Επιτροπή Γεωργίας, στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο. Το γεγονό ότι δεν πρέπει το στρατηγικό σχέδιο να υπηρετεί ειδικού στόχου των κρατών μελών, αλλά το ίστο όχι, θα πρέπει να ενταχθούν μέσα σε μια ευρύτερη και κοινή ε, γεωργική ευρωπαϊκή πολιτική. Επίσης η ανάπτυξη της υπαίθρου έχει πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερος όταν πρόκειται για τον προϋπολογισμό και τα ποσά που θα παραμένουν διαθέσιμα για τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα. Πρέπει επίσης να μιλήσουμε για επενδύσεις. Πιστεύουμε ότι οι επενδύσεις πρέπει να θεωρηθούν κομμάτι αυτής της υποστήριξης που θα προφέρουμε στη Γεωργία σε ορισμένες χώρες ε, που έχουν ε, μεγάλο ορεινό όγκο όπως η Βουλγαρία, αυτό θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πολύ σημαντικό το σχέδιο αυτό και πιστεύουμε ότι μπορεί να βρει άριστη εφαρμογή στη Βουλγαρία. Ω εκ τούτου έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία για τις περιοχές αυτές που είναι τόσο ευάλωτε. Σήμερα άκουσα ερωτήσεις σχετικές με συχνές πτωχεύσεις στον τομέα της γεωργίας. Ξέρουμε ότι οι αγορές είναι ανελέητες απέναντι στο γεωργό. Άρα πρέπει η γεωργική πολιτική να προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και γι' αυτό έχουμε και σχέδια χρηματοδότησης, επί παραδείγματι για την εκτροφή των ζώων. Ε, πράσινες πληρωμές επίσης είναι ένα άλλο ευαίσθητο θέμα. και σημαντικό μέτρο. Πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να διατηρήσουμε δηλαδή τον κανονισμό για την βιολογική γεωργία και ότι κάποια κράτη-μέλη φαίνεται να έχουν ε, κουραστεί πια από τις συζητήσεις εδώ και τρία χρόνια αυτού του κανονισμού. Ωστόσο εμείς φρονούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αποσταλεί ένα σαφές μήνυμα για τον προϋπολογισμό της ε, ΚΑΠ. Είναι πολλά τα τεχνικά ζητήματα που ακόμη δεν έχουν επιληθεί Πιστεύω πάντως ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για το τελικό αυτό έγγραφο για να ε, εγκριθεί. Επίσης, ε, οι εμπορικές πρακτικές. Ο θεμητός ανταγωνισμός είναι πολύ σημαντικό ε, θέμα. Θα αρχίσουμε από τις πρώτες μέρες να το συζητούμε. Άλλωστε πιστεύουμε ότι μέχρι τέλη Απριλίου ή τις αρχές Μαΐου θα έχει, λάβει, θα καταλάβει μεγάλο τμήμα της επικαιρότητα και του ενδιαφέροντος. Ε, πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι είναι σε διαστάσεις μικρότεροι, πιο ευάλωτοι, πιο αδύναμοι, που συχνά ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί δεν τους καταβάλουν τα δέοντα ή μεγάλη... Ε, οι μεγάλες επιχειρήσεις. Και ναι, μπορεί να υπάρχουν ε, συμβάσει, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν μερικοί αγοραστέ ή διαμεσολαβητέ, οι οποίοι ακόμη και συμβάσει δεν είναι διατεθειμένοι να υπογράψουν, που ούτω ή άλλω θα τηρούσαν. Βλέπουμε στη Βουλγαρία, παραδείγματι, συχνά γεωργοί να εργάζονται χωρί υπογεγραμμένη σύμβαση. Έρχονται, μα λένε, το δεν μου βγάλανε, και εμείς προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να κάνουν την καταγγελία στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχουν και ε, σώματα διαιτησίας για το χώρο αυτό. Σώματα διαιτησίας ή δικαστήρια βεβαίως ε, δεν συνεπάγονται απαραίτητα ότι τελειώνουν τα προβλήματα. Και έτσι περνώ στο θέμα της διανομής πόρων και εισοδημάτων, αναδιανομής πόρων και εισοδημάτων, μέσα σε όλη αυτή την αλυσίδα, αγοραστές ή διαμεσολαβητές, ε, παραγωγή, χρήστες, τελικός χρήστης, είναι, ε, ε, αποτελούν ένα σύστημα με πολύ λεπτή ισορροπία στην αγορά των γεωργικών προϊόντων. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα έτσι ώστε αυτή η συζήτηση να μην αναπαιμφθεί στο μέλλον, σε ένα μελλοντικό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις εκλογές. Εσωτερική αγορά, παρακολούθηση τιμών. Ξέρετε ότι πρόκειται για ε, ζήτημα αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει το παρατηρητήριο. Εμείς ωστόσο έχουμε ευθύνη να επιμείνουμε και να επιμένουμε τις ε, πληροφορίες και τα στοιχεία να τα ε, λαμβάνουμε τακτικά στα συμβούλια, έτσι ώστε να μπορούμε και να τοποθετούμαστε. Εσείς συγκεκριμένα αναφερθήκατε στη ζάχαρη. Ξέρουμε ότι υπάρχει ζήτημα και σε σχέση με το γάλα σκόνη, σε σκόνη. Και τα αποθέματα. Υπάρχει μια ιδέα, το γνωρίζουμε, για μια σταδιακή εξάλληψη των αποθεμάτων, ώστε να φτάσουν οι τιμές σε, μια, σε ένα σημείο ισορροπίας πιο ικανοποιητικό. Έχοντας εξετάσει τα στοιχεία του 2017, ε, μπορώ να επισήμανω ότι υπήρξε σταθερότητα τιμών και βελτίωση στις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στις ε, διεθνείς αλλά και τις ε, πολυμερείς και τις διμερείς διαπραγματεύσεις με διάφορες περιφέρειες του κόσμου και δίτη Μερκοσούρ. Βεβαίως έχουν πολιτικό σκέλος αυτές οι διαπραγματεύσεις. Οι τέσσερις χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν έχουν συμφωνία αντίστοιχη με τον υπόλοιπο κόσμο. Πρόκειται για μια σημαντική συμφωνία που τους επιτρέπει και μας επιτρέπει να αναπτύξουμε εμπορικές δραστηριότητες με τις χώρες αυτές και συναλλαγές. Πάντως ε, δεν πρέπει ποτέ να μου ότι εδώ διακυβεύεται το ίδιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Και ένα αμφίβολο. Πρέπει κάθε προϊόν που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρεί αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να υπάρχουν έλεγχοι. Ωστόσο, στον τομέα του βοήου κρέατος υπάρχει μεγάλος παραγωγός με προϊόν υψηλής ποιότητας που καθίσταται ανταγωνιστής, σκληρός και ξέρετε ότι πριν από δέκα μέρες ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες χωρίς, ε, πολύ ικανοποιητικό, χωρίς να δώσουν πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ε, κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να αντιπιστώσει κανεί και για τη συμφωνία με το Μεξικό. Για το λόγο αυτό το Συμβούλιο απαιτεί τακτικά η Επιτροπή να το ενημερώνει για τις συνομιλίες αυτές και ιδιαίτερα για τα βέστα αυτά θέματα τα οποία συζητούν τα κράτη-μέλη βέβαια. και όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Όντως πρέπει και αυτά να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό της γεωργικής πολιτικής, γιατί επηρεάζει βέβαια το κλίμα και το περιβάλλον η γεωργία, όπως άλλωστε μπορεί να συμβάλλει και σημαντικά στην διαφύλαξη των ε, φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος συνολικά. Εμεί θα θέλουμε να δούμε κάποιε λεπτομέρειε, να συζητήσουμε κάποιε λεπτομέρειε περισσότερο. Ε, μιλήσαμε για διάφορε συμφωνίε. Ο κ. και αναφέρθηκε συμφωνία με τη Ρωσία, το Ηνωμένο, στο, στο εμπορικό πόλο με τη Ρωσία. Ε, η Ουκρανία επίση αναφέρθηκε. Η κατάσταση με τη Ρωσία είναι τέτοια που ακόμη και αν ε, σταματήσει από πλευρά μα ε, ε, το εμπάργκο, η Ρωσία μάλλον δεν θα έχει ενδιαφέρον να προχωρήσει, διότι έχει κάνει τεράστιε επενδύσει σε πολλού τομεί. Και το να ανοίξουν τις αγορές μας, τις αγορές τους, σε ευρωπαϊκά προϊόντα πολύ καλής ποιότητας, θα σήμαινε απώλεια ε, του αναμενωμένου προϊόντος από τις επενδύσεις. Και αυτό αφορά βέβαια τις τράπεζες τους. Ξέρουμε ότι οι κυρώσεις ήχθησαν για λόγους άσετους με τη Γεωργία. Αλλά η Ρωσία έλαβε τις αποφάσεις της και εμείς στην Ευρώπη χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της υπερπαραγωγής. Κύριε Άγνιου, αναφερθήκατε σε πιθανές λύσεις. Όντως πρέπει να κεντρωθούμε στην καινοτομία. Και πιστεύω ότι κάποιες ε, πρακτικές στην ε, γεωργία επιτρέπουν τον περιορισμό των επιβλαβών ε, εκπομπών. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αγνοούμε τη σημασία της ασφάλειας των τροφίμων ή να παραγνωρίζουμε την ευαισθησία των πολιτών στο θέμα αυτό. Ταυτόχρονα η κτηνοτροφία και κυρίως των μερικαστικών έχει συνεπεί στο περιβάλλον. Και ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι αυτό της ευημερία των ζώων που ανέφεραν η κυρία Μίλλερ και άλλοι ομιλητές ε, με το παράδειγμα των μεταφορών. Οι υπηρεσίε της Ευρωπαϊκή Επιτροπής ελέγχουν τις σφαγές που λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνίες. Η Τουρκία είναι μία εξ αυτών. Αν όντω υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να ενημερωθούν οι αρχές σχετικά. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες ό,τι αφορά τη μεταφορά των ζώων προς την Τουρκία. Η Τουρκία ίδια είναι μια πολύ μεγάλη αγορά και κάνει και αναδιανομή των ζωικών προϊόντων και στον αραβικό κόσμο, στις χώρες του αραβικού κόσμου και γι' αυτό θεωρώ ότι τα ζώα δεν εξάγονται στην Τουρκία για να σφαγούν εκεί και να επανεισαχθεί το κρέας τους από την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το θέμα το συζητούμε συχνά με τις αρχές υγειονομικής υγείας των ζώων ε, στην Τουρκία και μάλιστα μιλούμε και για αυστηρούς ελέγχους ε, για τα ζανιοκτώνα, γιατί η ε, Τουρκία είναι πραγματικά μεγάλος εξαγωγός ε, φρούτων και λαχανικών προς την Ευρώπη. Και φυσικά στα σύνορα γίνονται πολλοί έλεγχοι. Προφανώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε 100% τα προϊόντα που έρχονται, αλλά παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τα συνοδευτικά έγγραφα και τα φορτία που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γίνει μια διάσκεψη για την ε, ευημερία των ζώων και για τις μεταφορές στις 24 Απριλίου, στη Σόφια συγκεκριμένα. Όλες οι αρχές που ασχολούνται με το θέμα αυτό βεβαίως θα είναι προσκεκλημένες. Τώρα, για την άγρια ζωή. Το συζητήσαμε και το πρωί. Θα γίνει μια διάσκεψη στη Βουλγαρία και νομίζω ότι και οι Πολωνοί συνάδελφοι θα κάνουν κάτι παρόμοιο την επόμενη εβδομάδα. Θα μελετήσουμε οριζόντια προβλήματα που προκύπτουν και πολλά από τα θέματα για, την, για τα ζώα που προκύπτουν ε, ας πούμε η αφρικανική πανόλη των χείρων που επηρεάζει κυρίως τα αγριογούρνα ή άλλες ε, επιζωτίες πτηνών. Πολύ συχνά ο φορέας της ασθένειας, της επιζωτίας, είναι κάποιο άγριο ζώο. Ας πούμε αποδημητικά πτηνά. Γι' αυτό πρέπει να μπαίνουν σε κάποια απομόνωση τα συγκεκριμένα ζώα όταν ε, τα ζώα εκτροφής όταν υπάρχει τέτοιος ε, κίνδυνος. Τον Ιούνιο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ένα σχέδιο για την ε, συνεκτικό για την ε, ευημερία των ζώων και βεβαίως τα κράτη-μέλη πρέπει να το εφαρμόσουν. Φυσικά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. γιατί υπάρχει και η, ε, το συνολικό πακέτο ε, για τα φάρμακα, τα κτηνιατρικά φάρμακα και την αντιμικροβιακή αντίσταση. Τώρα, η Βουλγαρική Προεδρία βεβαίως εκτιμά τις προσπάθειες που κάνει το Κοινοβούλιο και περιμένουμε και την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Τα σιτηρά υψηλής πρωτεΐνης είναι ουσιαστικά το 5% των, ε, της παραγωγής. Ο κύριος ε, ε, Νάικοφ ε, ανέφερε κάποια θέματα που αφορούν ε, αμυγός την, στη Βουλγαρία και βεβαίως μπορώ και διμερώς να τα συζητήσω μαζί του, αλλά όντως όλα αυτά που είπατε είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δεν δεν σας είπα να ολοκληρώσετε αμέσως, απλώς είπα να πλησιάζετε σιγά σιγά προς το τέλος. Μπορείτε να συνεχίσετε λίγο ακόμη, δεν ήθελα να σας διακόψω τόσο απότομα. Δεν ήθελα να ολοκληρώσετε έτσι ξαφνικά και απότομα, απλώς είπα να σιγά σιγά να πλησιάζετε προς το τέλος. Μπορείτε να συνεχίσετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει είπατε ότι δεν έχετε να προσθέσετε τίποτα άλλο, Ολοκληρώσετε την δευτερολογία σας. Και έκλεισε δυστυχώς το μικρόφωνο του Πρόεδρου. Υπάρχουν μήπως συμπληρωματικές ερωτήσεις. έχουμε την ευκαιρία για λίγο ακόμη ε, να παρατηρούμε τη συζήτηση, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες απορίες. Αφιερώσαμε σχεδόν δύο ώρες, μία ώρα και 50 λεπτά στην ανταλλαγή απόψεων με τον ε, Υπουργό Γεωργίας, που ήταν και ευρύτατη, κάλυψε ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων. Όσοι ζήτησαν το λόγο είχα την ευκαιρία να τον λάβουν και να μιλήσουν. Εκτενέστατη συζήτηση, οπότε αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις Η απορίες μπορούμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ευχόμαστε καλή επιτυχία κύριε Υπουργέ, καλή επιτυχία στη Βουλγαρική Προεδρία. Η δική σας επιτυχία θα είναι και για μας ε, επιτυχία, γιατί η στόχη μας είναι κοινή και θα είναι και κοινά τα επιτέγματά μας αν καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτούς τους ε, δύσκολους ε, στόχους. Πάντως ε, θα είναι ενδιαφέρουσα η Προεδρία σας και θα επηρεάσει ιδιαίτερο την μορφή της μελλοντικής κοινή γεωργικής πολιτικής. Και είναι φυσικό γιατί λαμβάνετε το λόγο σε μια εξαιρετική και πολύ δύσκολη στιγμή. Σας ευχαριστώ, λέει ο Υπουργός. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής σας για την ακρόαση αυτή, την ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ ε, για την προσοχή σας και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι από εδώ και πέρα και τους επόμενους μήνες και εγώ και το επιτελείο μου είμαστε στη διάθεσή σας. Ε, ξέχασα και μία ερώτηση, το ζήτημα του Brexit και την ερώτηση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Συμβούλιο δεν πρόκειται να πρωτοστατήσουμε στη συζήτηση. Το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας είναι περισσότερο μόνο για τα θέματα αυτά και όχι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά σας ευχαριστώ. Ε, ναι, σας ευχαριστούμε. Πραγματικά ήταν εκτενέστατη η ανταλλαγή απόψεων. Εντυπωσιακή. Κύριε κύριε Υπουργέ, ε, η, η ανταλλαγή απόψεων μαζί σας ε, συνέπεσε με άλλα δύο θέματα της ημερήσιας διάταξης, την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, της ειδική έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου για τον προγραμματισμό στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης και την λιγότερη πολυπλοκότητα και μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα. Ο κύριος Βοητσεχόφσκι θα μας κάνει την παρουσίαση της έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου και άλλο θέμα που θα πραγματευτούμε σήμερα είναι η πρώτη παρουσίαση της έκθεσης πρωτοβουλίας του κυρίου Ντόρφμαν σε σχέση με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ και καλή επιτυχία στη Βουλγαρική Προεδρία. If you, if you have uh, the logistic uh, problems, uh, tell me. Okay. I will organize everything. Thank you. Thank you. Thank you. Jak Państwo wiecie, wymiana poglądów była bardzo bogata. In, Όντως ήταν πολύ πλούσια αυτή η ανταλλαγή απόψεων και είχαμε και την ευκαιρία το πρωί από τις 8 να συναντήσουμε τον Υπουργό. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, το σημείο 12. Θα καλωσορίσω τον κύριο Βοητσεχόφσκι που ήταν παρόν και στην προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων και άκουσε την ομιλία του Υπουργού Γεωργίας της Βουλγαρίας. Ελάτε κύριε Βοητσεχόφσκι. Θα ασχοληθούμε εδώ με ένα πολύ σημαντικό θέμα και το γεγονό ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα διτέλεσε και αντιπρόεδρος της Επιτροπή Γεωργίας μας επέτρεψε να, να καταλήξουμε σε πολύ καλή γνώση των θεμάτων αυτών και σε πολύ εμπεριστατωμένη γνώση. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η παρουσίαση της ειδική έκθεσης ε, του ελεκτικού συνεδρίου γιατί αναφέρεται συχνά το θέμα των σχέσεων πρώτου και δεύτερου πυλώνα και τα όρια μεταξύ τους. Μετακή, μερικοί μιλούν μόνο για τον πρώτο πυλώνα, άλλοι μιλούν μόνο για τον δεύτερο πυλώνα. Και ο διαχωρισμός της κοινή πολιτικής σε δύο πυλώνες είναι πολύ σημαντικός και σίγουρα και στα πλαίσια της μεταρρύθμισης θα πρέπει να διαλευκάνουμε τις διαφορές τους. Θα σας δώσω τώρα το λόγο για την παρουσίαση της ειδική έκθεσης. Δυστυχώς επειδή σχεδόν δύο ώρες ε, μας πήρε το πρώτο θέμα, που ήταν βέβαια σημαντικό, αλλά μας έριξε λίγο πίσω, θα είμαι λίγο πιο αυστηρός και θα περικόψω κάπως το δικό σας ε, χρόνο. Παρακαλώ κύριε Βοητσεχόφσκι, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω εδώ την, ελπίζω, ενδιαφέρουσα και για σας, ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύθηκε πέρσι τον Νοέμβριο με τίτλο τον προγραμματισμό στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξη. Λιγότερη πολυπλοκότητα και μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα. Θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση αυτής της ειδική έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου και ελπίζω να είναι κατατοπιστική. Καταρχήν όλοι γνωρίζουμε εδώ πόσο σημαντική είναι η αγροτική ανάπτυξη και το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ε, που είναι εφοδιασμένο περίπου με 100 δισεκατομμύρια ευρώ για μια επταετία περίπου 15 δισεκατομμύρια το χρόνο και βλέπετε εδώ σε σύγκριση με την αγροτική ανάπτυξη ε, τη σύγκριση μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Ε, το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει περίπου 50 δις μερίδιο. Τώρα, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι των κονδύλιων της αγροτική ανάπτυξη. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Πολωνία, η Ισπανία και η Ρουμανία. Αυτή είναι οι σημαντικότεροι παραλήπτε των κονδύλιων της αγροτική ανάπτυξη. Η διαδικασία του προγραμματισμού οργανώνεται σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο σε μερικές χώρες μέλη. Και θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι ο σωστός προγραμματισμός είναι το κλειδί της επιτυχίας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Εμείς εξετάσαμε και ελέγξαμε 12 από ε, τα 118 προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Αυτός είναι ο συνολικός αριθμός ε, των ε, προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 118 είναι συνολικά. Εμείς ελέγξαμε 12 από αυτά. Το πολωνικό, ρουμανικό, ε, ελληνικό, ιταλικό από την Καμπανία, αυστριακό, ε, του, της Βάδης Βιντεβέργης του κρατηδίου από τη Γερμανία, της Λορένης στη Γαλλία, της Βαλονίας στο Βέλγιο, το Ιρλανδικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και με όχι άμεσα, αλλά με υλικό τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ελέγξαμε και τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης Αγγλίας και της Δανία. ξέχασα και το πρόγραμμα της Λαριόχα, της περιοχής Ριόχα της Ισπανίας. Ποιες ήταν οι ερωτήσεις που θέσαμε στον έλεγχο. Ε, το νομοθετικό πλαίσιο αντικατοπτρίζει την ε, έμφαση στην ε, επίδοση Πώ συμβάλλουν τα προγράμματα αγροτική ανάπτυξη στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και πώ θα χειρίζεται τον προγραμματισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ποια ήταν τα βασικά συμπεράσματα αυτή τη ειδική έκθεση. Τα συμπεράσματα μα είναι ότι τα προγράμματα αγροτική ανάπτυξη παρά είναι γενικά, ε, υπερβολικά μακροσκελή και περίπλοκα, η διαδικασία προγραμματισμού υπερβολικά μακροπρόθεσμη και μάλιστα ε, πολύ καθυστερημένα εγκρίνονται μερικά αγροτικά προγράμματα, προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και ελάχιστα προσανατολίζονται στα αποτελέσματα. Υπερβολικά γενικά, λοιπόν, αυτό ήταν το... η πρώτη αιτίαση. Οι ανάγκες ε, περιγράφονται πολύ γενικά και αόριστα. Τα μέτρα επικεντρώνονται στις δράσεις και όχι στα αποτελέσματα και ήταν δύσκολη η εκτίμηση, η αξιολόγηση του κατά πόσο οι ανάγκες ε, ικανοποιούνται από τη λήψη των μέτρων. Εμείς ε, ενδεικτικά σας λέω, γιατί δεν ασκούμε κριτική στα κράτη-μέλη, είναι παραδείγματα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και εντοπίσαμε σε όλα τα προγράμματα που ελέγξαμε. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, να αυξήσει και να διαφοροποιήσει τον αριθμό των θέσεων εργασία στην, στην Ήπεθρο. Πολύ γενικέ αυτέ οι ανάγκε και όριστες. Δεν γίνεται σωστή περιγραφή. Το πολωνικό πρόγραμμα μιλάει για αποκατάσταση και διαφύλαξη της βιοπικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης και της Natura 2000 σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το περιβάλλον. Και στην Ιρλανδία ένα καλά στοχοθετημένο και προγραμματισμένο πρόγραμμα αγροπεριβαλλοντικό. Ωραία όλα αυτά, αλλά παρά είναι γενικά και αόριστα. Και εδώ έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που δείχνει ότι παρά είναι περίπλοκα και μακροσκελή τα έγγραφα. Εγώ θυμάμαι ότι ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας ε, ως Ευρωβουλευτής ε, συμμετείχα στη συζήτηση που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γεωργίας θα πρέπει να απλοποιηθεί. Εδώ συγκρίνουμε τον αριθμό των σελίδων, ε, την τεκμηρίωση αυτών των προγραμμάτων στην ε, δημοσιονομική περίοδο 2007-2013, στην προηγούμενη δηλαδή περίοδο προγραμματισμού και στην τρέχουσα περίοδο 2014-2020. Διαπιστώνουμε δηλαδή έτσι ότι σε όλα τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης έχουμε διπλάσιο αριθμό εγγράφων και σελίδων από ό,τι στο παρελθόν. Με μία μόνο εξαίρεση την Ιρλανδία το Ιρλανδικό πρόγραμμα είναι το ε, συντομότερο και μάλιστα και μία σελίδα συντομότερο από το προηγούμενο, της προηγούμενης περίοδου προγραμματισμού. Τα περισσότερα πάντως προγράμματα ήταν διπλάσια από την προηγούμενη περίοδο. Στην Ιταλία, στην Καμπανία, το πρόγραμμα αργοτικής ανάπτυξης στην προηγούμενη περίοδο 2007-2013 ήταν 422 σελίδες και στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού είναι πάνω από 1000 σελίδες. Και σε άλλα κρατημέλη το ίδιο παρατηρούμε. Με εξαίρεση επαναλαμβάνω την Ιρλανδία που είχαμε μία σελίδα λιγότερη στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Εμείς ε, παρατηρήσαμε ότι είναι υπερβολικά απαιτητική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες που εκπονούν τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Είναι πολλά αυτά που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια τα προγράμματα βρίθουν ε, ε, ενδιαφέρον των στοιχείων, αλλά τα στοιχεία αυτά είναι ενδιαφέροντα για τους ακαδημαϊκούς, για τους πανεπιστημιακούς, όχι για τους γιαουργούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παρά είναι πολλά τα στοιχεία που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ βλέπετε σε μια άλλη απεικόνηση με το ίδιο πρόβλημα. Επίσης, εμείς συστήνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλούστευση του περιεχομένου των προγραμμάτων και μείωση του αριθμού των απαιτήσεων, των προϋποθέσεων των απαιτουμένων. Αυτή είναι η σημαντική σύσταση. Απλούστευση και συντόμευση των προγραμμάτων. Άλλο θέμα. Η περίοδος προγραμματισμού παρά ήταν μακροπρόθεσμη, εκτινόταν σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Βλέπετε στη φωτογραφία αυτή πόσο διήρκησε η έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Από τη στιγμή που υπευλήθη το πρώτο σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το κράτος μέλος ή από την αρμόδια περιφέρεια, πέρασε σχεδόν ένας χρόνος, 11,5 μήνες. Αυτό είναι ο μέσο όρο τη διάρκεια τη διαδικασία. Σε μερικέ χώρε είναι λίγο συντομότερο το διάστημα αυτό, αλλά είναι σχεδόν ένα χρόνο ε, υπερβολικά χρονοβόρα διαδικασία. Και πολύ σημαντική αυτή, αυτή η εικόνα, αυτός ο πίνακας που συγκρίνει τη διαδικασία της έγκρισης των προγραμμάτων ε, αγροτικής ανάπτυξης στην περίοδο 2007-2013 την νομοθετική διαδικασία που ξεκίνησε το 2004 και όλα ήταν έτοιμα ήδη στις αρχές του 2007. Ενώ στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού η έγκριση του εφαρμοστικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Περιοχής έγινε το 2014, τον Ιούλιο του 2014, έξι μήνες δηλαδή μετά την έναρξη της δημοσιονομικής περίοδου. Υπερβολικά αργά δηλαδή. Και μια άλλη σημαντική πληροφορία. Εδώ συγκρίναμε τις δαπάνες του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ανάπτυξης ε, Αγροτικής Ανάπτυξης στο τέλος της ε, ε, περίοδου προγραμματισμού. Στην πρώτη περίοδο 2007-2013, κατά τα τέλη ε, το 2010, τέλη του 2010, μετά από τέσσερα χρόνια, ε, το 29% των κονδύλιων είχαν δαπανηθεί και το 71% των κονδύλιων δεν είχαν ακόμη δαπανηθεί, δεν είχαν εκταμιευθεί. Στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού ε, βρισκόμαστε στα τέλη του 2017 και μόνο το 21% των κονδύλιων έχουν δαπανηθεί και το 79% των κονδύλιων παραμένουν αχρησιμοποίητα. Εδώ σας παρουσιάζουμε το ρυθμό απορρόφηση εκταμίευση ε, των κονδυλίων του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στα τέλη του 2010 σε σύγκριση με τις δημοσιονομικές προοπτικές. Στα τέλη του 2010 λοιπόν, μετά από τέσσερα χρόνια εφαρμογής ε, της δημοσιονομικής περίοδου, δύο κράτη-μέλη είχαν πάνω από 50% απορρόφηση. Η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο τότε ήταν τα κράτη με τον καλύτερο ρυθμό απορρόφησης. Ε, και κανένα κράτος δεν ήταν κάτω από 15% ρυθμό απορρόφησης. Τώρα, εν έτη 2017 δεν έχουμε ούτε μία χώρα πάνω από 15%. Πάνω από 50% μάλλον. Η Φιλανδία είναι στο 43% και η Ιρλανδία ένα υψηλό ποσοστό. Αλλά ούτε μία χώρα δεν είναι πάνω από το 50%. Θυμάστε ότι στην Ιρλανδία είχαμε το συντομότερο πρόγραμμα αγροτική ανάπτυξη. και επίση είναι σε δεύτερη θέση ό,τι αφορά το βαθμό απορρόφησης. Δεν έχουμε εδώ καμία ταξινόμηση, μια εικόνα. Αλλά έχουμε έξι κράτη-μέλη στα οποία ο ρυθμός απορρόφησης είναι κάτω του 15%. Κάτι που δεν συνέβαινε στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Ποιε ήταν οι συστάσει μα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συστήνουμε την έγκαιρη υποβολή των νομοθετικών προτάσεων για την αγροτική ανάπτυξη ε, μετά το 2020, ώστε να γίνει εμπρόθεσμα η έναρξη στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Και ποια είναι τα συμπεράσματα μετά τα προβλήματα που εντοπίσαμε. Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης δεν ήταν επαρκώς ε, προσανατολισμένα στα αποτελέσματα και ένα καλό παράδειγμα αυτού του προβλήματος είναι οι πίνακες που σας έδειξα και θυμάστε την ε, ειδική έκθεση για τους νέους γεωργούς που σας παρουσίασα τον Ιούλιο. Οι νέοι αγρότες ε, έλαβαν στην περίοδο 2007-2013 από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ, 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τους νέους αγρότες στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού και τα αποτελέσματα είναι στον κάτω πίνακα όπου βλέπουμε το ποσοστό μείωσης του αριθμού των νέων αγροτών στα κράτη-μέλη. Με εξαίρεση δύο κράτη-μέλη, τη Σλοβενία και τη Ρουμανία, όπου είχαμε αύξηση του αριθμού των ε, νέων αγροτών. Στα υπόλοιπα κρατημέλη, παντού αλλού, ο αριθμός των, ε, ο αριθμός των νέων γεωργών μειώθηκε, των νεαρών γεωργών μειώθηκε. Το ίδιο και με τις αγροτικές εκτάσεις. Οι αγροτικές εκτάσεις, ε, δηλαδή ο αριθμός των εκταρίων που χρησιμοποιούν οι νέοι γεωργοί, μειώθηκε από 57,7 το 2005 σε 51,9 το 2013. Οπότε δεν έχουμε ηλικιακή ανανέωση, ούτε και αποτελεσμάτα εντυπωσιακά από την μεγάλη υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων προς συνέρους Γιώργους. Και αυτός ο πίνακας δείχνει τα προβλήματα που έχουμε. Ότι μόνο δύο κράτη-μέλη δηλαδή παρουσιάζουν ποσοστό νέων γεωργών πάνω από 10%. Δηλαδή μιλούμε για γεωργούς κάτω των 35. Μόνο η Αυστρία και η Πολωνία έχουν πάνω, πάνω από 10%. Και σε τρεις χώρες έχουμε τους πιο ηλικιωμένους γεωργούς. Άνω των 65 ετών. Βέβαια είναι κάτω το 10% η Γερμανία, Αυστρία και Πολωνία. Και το 1 τρίτο των ε, Ευρωπαίων αγροτών είναι άνω των 65. Μόνο σε τρεις χώρες το ποσοστό τους ήταν κάτω των, 10%. Βλέπετε από τους πίνακες αυτές τα προβλήματα, τις πρακτικές συνέπειες του προγραμματισμού και τα αποτελέσματα. Και σας παρουσιάζουμε εδώ δύο παραδείγματα, ένα από την Πολωνία και ένα από την Ιταλία. Και πάλι δεν είναι κριτική προς τα κράτη-μέλη. Ε, το πρόβλημα δεν είναι τα κράτη-μέλη, το πρόβλημα είναι ο τρόπος της υποστήριξης. Στην Πολωνία ένας νέος δικαιούχος ε, είχε μια εκμετάλλευση 513 εκταρίων και έλαβε 100.000 ευρώ το χρόνο άμεσες ενισχύσεις και επιπλέον 3.000 ευρώ ως νέος γεωργός. Ποια, ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτής της ενίσχυσης για την ηλικιακή ανανέωση. Κανένας αντίκτυπος δεν υπάρχει. Καμία σχέση μεταξύ της βοήθειας, της ενίσχυσης και της ηλικιακής ανανέωσης στην Πολωνία. Δεύτερο παράδειγμα από την Ιταλία. Είχαμε μια εταιρεία που έλαβε την ενίσχυση του νεαρού Γεωργού, γιατί ένας από τους μετόχους είχε 16% ε, μερίδιο στην εταιρεία και χάρη σε αυτή την παρουσία η εταιρεία έλαβε 8.000 ευρώ το 2016 ενίσχυση. Η συνέπεια για την ηλικιακή ανανέωση, καμία απολύτως στις δύο αυτές περιπτώσεις. Και τέλος θα ήθελα να σας πω ότι φέτος το Μάρτιο θα ετοιμάσουμε ένα σύντομο έγγραφο προβληματισμού ως προς τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αυτό το έγγραφο προβληματισμού θα περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις μας ε, για τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, παρατηρήσεις που θα στηρίζονται στις ε, εκθέσεις μας, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις μας. Πάντως, δυστυχώς, έχουμε πολύ ανησυχητικά, τραγικά στοιχεία στις εκθέσεις μας. Την τελευταία δεκαετία έχουμε χάσει 4 εκατομμύρια αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Χάσαμε περίπου 20 εκατομμύρια εκτάρια γεωργικών γεών. Περίπου 20 εκατομμύρια εκτάρια γεωργικής γης χάθηκαν. Έχουμε πρόβλημα με τη Γύραση του γεωργικού πληθυσμού, δεν υπάρχει επαρκή ηλικιακή ανανέωση και έχουμε και πρόβλημα με την υπερβολική περιπλοκότητα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση των πολιτικών ηθινόντων και των πολιτικών ειδικά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει οι πολιτικοί ηθινόντες να βρουν μια λύση για να απλουστεύσουν την κοινή γεωργική πολιτική και να τη βελτιώσουν στο μέλλον. Το είπα και στην παρουσία της ειδικής έκθεσης για τους νέους αγρότες. Το επαναλαμβάνω και σήμερα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαμορφώσουμε μια νέα κοινή γεωρική πολιτική με διορατικότητα, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, όχι επταετή ορίζοντα, κοντόφθαλμο, αλλά για 27 ετή ορίζοντα πολύ πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα και θα πρέπει από τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και ίσως είναι καλή στιγμή η Βουλγαρική Προεδρία για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Πώς θα σχεδιάσουμε την κοινή γεωργική πολιτική με μία διορατικότητα, με μία μακροπρόθεσμη προοπτική και ποιες είναι οι προσδοκίες μας από το μέλλον της Γεωργίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Βοτσεχόφσκι. Έχουμε την ειδική αυτή έκθεση μεταφρασμένη σε όλες τις γλώσσες, επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και είναι προσβάσιμη αυτή η έκθεση. Οπότε παρακαλώ να περιοριστείτε σε ερωτήσεις ή σχόλια που δεν θα ξεπερνούν όμως το λεπτό. Να με συμπαθάτε για τον περιορισμό, αλλά επεκταθήκαμε υπερβολικά στην προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων με τον εκπρόσωπο της Βουλγαρικής Προεδρίας. Τώρα θα περιοριστούμε. Ο κύριος Ουαζό. Ένα λεπτό παρακαλώ, μόνο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, του Περιφερειακού Ταμείου, μάλλον το έχουμε δει. Εγώ είμαι εκπρόσωπο σε περιφερειακό επίπεδο, δεν έχει φέρει τίποτα το θετικό. Ε, ενώ θα έπρεπε να μειώνει την φτώχεια δίκτυου, υπηρεσία δικτύου, με συνέπειε και για τι επιχειρήσει και για του πολίτε. Τι συνέπειε νομίζω μπορεί να τι δει ο καθένα. σω θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχω αυτά τα καθήκοντα, δεν με έχει πλησιάσει κανεί. Ευχαριστώ κύριο Σανδρίο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομο. Ευχαριστώ καταρχάς το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για την έκθεση αυτή που έρχεται τη στιγμή που έγινε γνωστή και ανακοίνωση Επιτροπής. Θα αποβεί πολύ χρήσιμη αυτή η ενημέρωση. Δείχνει άλλωστε και τη βούληση των επιτρόπων, του επιτρόπου να προχωρήσει προ στόχου αυτού, αλλά ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ότι δεν έχει εφεύρει και τίποτα το κενό. Υπάρχουν συγκεκριμένα όρια, αυτό είναι όλο, με γνωστέ διαδικασίε. Άρα πρέπει να προσδιοριστεί το επίπεδο των στόχων μέσα στι γνωστέ διαδικασίε. Και πρέπει να είμαστε θέση ποσοτικά αλλά και ποιοτικά να αξιολογούμε τι δράσει. Και γι' αυτό χρειάζεται προσδιορισμό των στόχων, του επίπεδου των στόχων. Αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να γίνει. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξή. Γιατί δεν προβήκατε σε αξιολόγηση του Λίντερ στις διάφορες περιφέρειες. Εδώ τίθεται το ζήτημα της συνοχής ε, των περιοχών μεταξύ τους. Εδώ νομίζω ότι η καταγραφή της εδαφική συνοχής για τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους θα έχει πολύ μεγάλη σημασία και επίσης, ευχαριστώ σας βέβαια για τις καταλεκτικές παρατήρησεις ως προς τη δυνατότητα για σχεδιασμό μιας ε, ε, ολιστικής πολιτικής βράχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα και όχι βράχυπρόθεσμο σχεδιασμό. Ευχαριστώ κύριε για τη χρηματοδότηση. Δεν συμβάλλουμε στην επιδείνωση της κατάστασης για τις περιφέρειες που θα δυνατούν πια να τηρήσουν τα προγράμματα. Δεύτερη ερώτηση. Ζητάτε και τις επανεθνικοποίησεις Επίση, προθεσμίε. Σίγουρα να δώσουμε πρώτα λύση στην αγροτική ανάπτυξη πριν προβούμε σε μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική. Δεν είναι άδικο να μα. Πολύ και συγχαρητήρια για τα αγγλικά σας που βελτιώθηκαν άρδιν από τότε που σας έχω γνωρίσει. Τεράστιο επίτευγμα, πόσο δε μάλλον η σας είναι ήδη πολύ δύσκολο. Και ευχαριστώ πολύ και για την έκθεση από το ελεγκτικό συνέδριο. Πυρσός ελπίδας να μας επισέσματα καθυστερήσεις, δεν υπάρχει αξιολόγηση των επιδόσεων, υπερβολική πίεση στους δικαιούχους, ε, πιέζονται οι δικαιούχοι, οι ετούντες να ε, καταθέσουν με ασφικτικές προθέσεις. Τι πήγε αριστερά. Κύριος δυνανό. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ ιδιαίτερα για διαφορετικέ ερμηνείε. Όταν είχα εγώ καθήκοντα σε τοπικό επίπεδο, διαρκώ καταριόμουν τι διαδικασίε αυτέ, γιατί πάντα αισθανόμουν ότι ήμουν ο κακό μαθητή και έχω έναν αυστηρό δάσκαλο που στην απόγνωση το χώρο τη υπαίθρου. Μακάρ... Κάρθη. Ο ελεγκτικό συνέδριο θα κάνει κάποια ε, αναχώρα ε, έρευνα γιατί για την Ιρλανδία είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Τα 10,5 εκατομμύρια ε, και πραγματικά είναι πολύ ανησυχητικό το ποσοστό. Το Λίντερ στράφηκε. Οι δικές σας οι προτάσεις ε, παλαιότερα χρησιμοποιούνται ως αιτιολόγηση για το γιατί συνέβη αυτό και γιατί δεν έχει υπάρξει συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Οπότε παρακαλώ θα κάνετε κάποιο είδους τέτοια έρευνα αναχώρα συγκεκριμένη για το πόσο, πώς αντί να... Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας. Ένα σημείο θέλω να τονίσω. Η ε, ενίσχυση των ε, ε, νέων ε, δραστηριότητά του. Και επίσης, μιλήσατε για την αλλαγή των γενεών που δεν πάει όπως θα έπρεπε, αλλά νομίζω ότι και για αυτό όταν ανικώς αποδεκτό το επάγγελμα του Γιώργου Βεβαίω πρέπει να λάβουμε υπόψη και όλα τα υπόλοιπα θέματα τη προστασία των ζώων. Ευχαριστώ. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα παρούσα σε μια αντίστοιχη ε, συνάντηση που είχε να κάνει κυρίω με την παρουσίαση των αριθμητικών που έχουμε ψηφίσει, που έχουμε συμφωνήσει κατά πόσο το έχετε μελετήσει, αν ε, θεωρείτε ότι πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση, γιατί για μας είναι σημαντικό που λαμβάνουμε τις πολιτικές αποφάσεις, να δούμε και τι θα, πώς θα προχωρήσουμε στη συζήτηση για την κοινή αγροτική πολιτική. Και επίσης πρέπει να ρίξουμε και μια ματιά στα περιφερειακά προγράμματα κομισιών να αφήσει δηλαδή περιθώριο στις, ε, ελιγμών στις περιφέρειες. Πώς μπορούμε να τα, κατα, να τα καταφέρουμε χωρίς όμως να αυξήσουμε την, ε, το διοικητικό άχθος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ροπέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την παρουσίαση αυτή. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα για μας. Πρέπει να αναλάβουμε δράση στον τομέα αυτό. Αρκετά μιλάμε για τα προβλήματα και θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Είπατε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της προγραμματικής περίοδου υπήρξε μια καθυστέρηση ενός εξαμένου ε, περίπου σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Τα κράτη-μέλη είχαν προετοιμάσει μακροσκελέστερα κείμενα, θέλανε να συμπεριλάβουν και άλλα στοιχεία. Η καθυστέρηση αυτή είχε να κάνει με τις νέες απαιτήσει που ίσως προέκυψαν και δεν ήταν γνωστές εγκαίρως. Αν τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβάνουν πολλά στα προγράμματά τους, πολλά στοιχεία, τότε ίσως θα μπορούσαμε να περιορίσουμε λίγο τις απαιτήσει. Και επίσης να θέσω και ένα ίσως ρητορικό ερώτημα. Μιλούμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι ε, γεωργοί, ε, οι ε, πιο μεγάλες ηλικίε γεωργοί, τα, τα τρόφιμα πότε θα αρχίσουν να μας λείπουν. Η ε, κυρία Πετήρ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και καλωσορίζω τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ο ρυθμός απορρόφηση των κρατών μελών είναι 21,4%. 12 κράτη-μέλη βρίσκονται κάτω από αυτό το μέσο όρο το που στένουν, ε, ενώ κονδύλια υπάρχουν και δεν εκταμιεύονται. Ο κύριος Μπούντα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ λακωνικός έχουμε υποβάλει το φάκελό του ένας Γιώργος. Ε, δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να προβλέψουμε ενοποιημένε και απλουστευμένε διαδικασίε σε όλα τα κράτη κονδυλίων, αλλά πώ να βελτιώνεται ο αριθμό εκταμείευση, αν είναι τόσο περίπλοκε οι διαδικασίε. Ναι, αλλά τα λεφτά είναι λεφτά. Κύριε Κάντεμπαχ. Του τελευταίου μήνε και δύο χρόνια είναι πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο οδηγίες χρήσεως, ιδιαίτερα δεδομένου ότι θα έχουμε λιγότερα κονδύλια από ό,τι αναμένεται στο μέλλον και λόγω του Brexit αλλά και λόγω ε, της αύξησης των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με την ασφάλεια, με το μεταναστευτικό κτλ. Ε, καλό θα είναι λοιπόν να μην χάνονται, να μην γίνονται οι περικοπές και οι εξοικονομήσεις εκεί που δεν πρέπει να γίνονται στο λάθος σημείο. Τα κονδύλια λοιπόν που δαπανώνται θα πρέπει να προσφέρουν την προσθεμένη αξία, την ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία, να δίνουν κίνητρα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και κυρίως ε, με το βλέμμα στρεμμένο σε μια νέα ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική. Πρέπει να κάνουμε επιλεκτικές παρεμβάσεις και όχι με την μπουλντόζα να περικόψουμε κατά 50%. Αν είστε και εσείς αρκετά επιγραμματικοί. Κυρία Λουίς Χόφμαν. Okay, yeah, I think that's better. So thanks very much. Έκθεση. Η ουσία τώρα των συστάσεων αυτών ε, βεβαίω ε, είναι σημαντική, τις δεχόμαστε, κυρίως γιατί συμμεριζόμαστε και εμείς την άποψη ότι για πολλούς, ε, σε πολλούς τομεί είναι δυνατόν να γίνουν βελτιώσεις. Τους τομείς του οποίου για το μέλλον της Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να επιτύχουμε ένα καλύτερο πλαίσιο, πιο απτό για την παροχή των ενισχύσεων. Βεβαίω η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη. Ξέρουμε ότι πρέπει να πλουστεύσουμε τα πράγματα, πρέπει να βρούμε πιο απλούς τρόπους. Τρόπους όμως. Τώρα, για κάποια από τα θέματα που αναφέρθηκαν. Ένα εξ αυτών είναι το θέμα της καθυστέρησης και η διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων. η διαδικασία συνολικά, από την αρχή δηλαδή, τη στιγμή δηλαδή που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή της, μέχρι την έγκριση της ε, βασικής πράξης, που πήρε 12 μήνες περισσότερο από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Ε, είμαστε σε διαδικασία συναπόφασης. Τώρα, από τη στιγμή που έχει εγκριθεί η βασική πράξη μέχρι να εγκριθεί και το τελευταίο καθυστέρηση ως την εξέβριση της νομικής βάσης, και την έγκριση αυτής. Από εκεί και μετά ε, ε, μπορέσαμε να ζητμίσουμε την περίοδο και πολύ πιο σύντομα να εγκρίνουμε τα ε, προγράμματα. Το άλλο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι το θέμα του επίπεδο δαπανών. Όντως, σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο υπάρχει μια μικρή μείωση ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε ακόμη επιτύχει τα όσα είχαμε επιτύχει στην αντίστοιχη περίοδο της περσινής χρονιάς. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω είναι ότι το Ταμείο άλλα κονδύλια, δηλαδή Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ταμείο Συνοχής και Κοινωνικό Ταμείο, είναι στο 8%. Οπότε νομίζω με τα άλλα ταμεία. Είμαστε περίπου τρία, τρεις φορές παραπάνω από τις ε, δαπάνες που έχουν τα άλλα ταμεία. Και επίσης ε, εδώ βρισκόμαστε αυτή τη, στιγμή, αυτή τη στιγμή σε σχέση με την εκτέλεση των κονδύλιων. Τώρα, εμείς είμαστε το μόνο δομείο που έχουμε δείκτες που επιτρέπει μέτρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των αποτελεσμάτων. Επίσης, υπήρχαν και κάποια άλλα σχόλια. Την τελευταία περίοδο δεν χάσαμε ε, επιφάνεια γεωργική. Τα 20 εκατομμύρια πούμε, εκτάρια που κάπου χάθηκαν από διεδαφών εκτάσεων από τα στοιχεία μας. Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη που σας περιόρισα. Γιάννους Βοητσεχόφσκι, έχει το λόγο. Χρόνου φίδου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και τη θετική σας ε, γνώμη για την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Σε ό,τι φορά την τελευταία πληροφορία που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η οικολογικοποίηση που δημοσιεύθηκε πριν τρεις μήνες και ήταν στοιχεία που δεν αφισβητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και οι γεωργικές εκτάσεις ήταν τότε 164 εκατομμύρια εκτάρια το 2005 ενώ το 2010 εκτάρια και μάλιστα υποβάλαμε αυτά τα στοιχεία στην προηγούμενη μας έκθεση για την οικολογικοποίηση και δεν αφισβητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, εμείς δεν επικρίνουμε τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες που εκπονούν τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπερβολικά απαιτητική. Ζητά πάρα πολλά από τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Θα πρέπει να πλουστεύσει οπωσδήποτε τα απαιτούμενα τις προϋποθέσεις που ζητά, που είναι υπερβολικές. Και αυτό θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και στην ε, επόμενη ΚΑΠ θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλούστερες ρυθμίσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιο απλά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Και ήταν ο έλεγχος της διαδικασίας προγραμματισμού και όχι των προγραμμάτων, γιατί το leader ήταν πρόγραμμα και όχι διαδικασία προς τους κυρίους Φλάνακαλ και Κάρθη. Και μάλιστα αύριο θα παρουσιάσω τη συγκεκριμένη ειδική έκθεση στην Ιρλανδική Βουλή, στην Επιτροπή Γεωργίας της Ιρλανδικής Βουλής. Οπότε αν μου επισημάνουν κάποια προβλήματα του προγράμματος Leader, θα προτείνω και εγώ να επανέλθουμε σε μελλοντικό έλεγχο και στο πρόγραμμα Leader. Δημιουργεί η πολύ καθυστερημένη έγκριση του προγράμματος. Τώρα ξεκινάμε τη συζήτηση γιατί μέχρι στιγμής μόνο 20-21% των κονδύλιων έχουν εκταμιευθεί μέχρι στιγμής. Και δεν είναι αρκετό αυτό το ποσοστό για να αξιολογήσουμε την αποτέλεσμα δημοσιονομικού. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το αριθμό εκτέλεσης της προηγούμενης περίοδου προγραμματισμού. Α, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε κύριε Βοητσεχόφσκι. Πολύ χρήσιμη η έκθεσή σας. Και Καλό κουράγιο, όπως λέμε, και στις μελλοντικές σας εργασίες. Μπορείτε να παραμείνετε. Επίσης, είχαμε μια συνεδρίαση για το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής. Ο κ. Ντόρφμαν, που θα συνοψίσει την θέση της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε λίγο χρόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της ΚΑΠ και χαίρομαι που ανέλαβα εγώ ως εισηγητής την αρθούνη νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό σκόπιμο θα ήταν το αργότερο στην Ολομέλεια του Ιουνίου ε, ε, δύο λόγια τώρα επί της αν δει κανεί την έκθεση του Επιτρόπου, η βασική αρχή είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της κοινή. Υπάρχουν νέε προκλήσει που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως το θέμα τη ε, ενισχυμένη βιωσιμότητα, ε, η ε, αλλαγή του περιβάλλοντο, Υπάρχουν νέε προκλήσει που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως το θέμα τη ενισχυμένη βιωσιμότητα, η αλλαγή του περιβάλλοντο που έχουμε και συζητούμε από την προηγούμενη μεταρρύθμιση. καθώς επίσης και οι διάφορες ε, συμφωνίες η ενισχυμένη επικουρικότητα. Ε, προσωπικά πιστεύω ότι σε κάποιους τομείς αυτό είναι σκόπιμο να υπάρξει, ας πούμε για τους ελέγχους ή αν δούμε κάποιους τομείς του προγραμματισμού. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μόνο μέσω της επικουρικότητας δεν θα υπάρξει απλούστευση για το χρονοδιάγραμμα αυτό. Αν ε, το δούμε αυτό, θεωρώ ότι ο πρώτος ε, πυλώνας να ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο, αλλά ο ε, δεύτερος ε, ρυθμίζεται και μερικός εθνικός, μερικός ευρωπαϊκός. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Θα συμπτύξουμε ίσως, δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να τα εμπλέξουμε, αλλά δεν θέλουμε σίγουρα να υπάρξει περαιτέρω διοικητικό αυτός. Και αυτό που σίγουρα πρέπει να αποφύγουμε είναι αυτή η επικουρικότητα που θέλουμε, η ενισχυμένη επικουρικότητα, το σύνολο της ε, κοινωνικής αγροτική ε, πολιτικής ε, να το προστατεύονται ας πούμε περισσότερο από γεωργούς που βρίσκονται σε χώρες οι οποίες δεν έχουν τόσο ανεπτυγμένα συστήματα. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ε, προστατεύονται ας πούμε περισσότερο ε, από γεωργούς που βρίσκονται σε χώρες οι οποίες δεν έχουν τόσο ανεπτυγμένα ε, συστήματα. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν καλύτερη ή σημανό πρόσβαση σε ό, στα κονδύλια για όλους τους γεωργούς. Επίσης ενδιαφέρον είναι το θέμα του ξεκαθαρίσματος, ότι αφήνει πριν από ένα χρόνο στην, στα πλαίσια της έκθεσης DES για την προετοιμασία των τρεχών των κανόνων, πρέπει να πούμε ότι πολλά συμπεριλαμβάνονται ήδη. Υπάρχει δηλαδή μια καλή βάση διασταυρούμενης συμμόρφωσης, υπάρχει ε, ένα φάσμα διαφόρων κανόνων βιωσιμότητας. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον τομέα της ε, ε, ανάπτυξης υπαίθρου κυρίως εκεί που υπάρχουν κοινό οργανώσεις αγοράς, να παραμείνουν και ίσως και να ενισχυθούν. Και τα τελευταία χρόνια είδαμε να προκύπτουν ε, συχνά έκτακτες καταστάσεις και κρίση για την ε, διαχείριση του κινδύνου. Υπάρχουν κάποια στοιχεία και νομίζω ότι στα πλαίσια του Omnibus έχουν ληφθεί κάποιε σχετικέ αποφάσει. Δεν νομίζω ότι στα πλαίσια τη ε, διαχείριση του κινδύνου δυνάμει του Omnibus θα καταλήξουμε ή θα χρειαστεί να κάνουμε τίποτα καινούριο. Νομίζω ότι αρκεί αυτό που ήδη έχει συμφωνηθεί. Οπότε οι εισηγητέ. Αυτά από μένα και ευχαριστώ το τον κύριο Λάιον. Μερικοί θα τον θυμούνται. Θα θυμούνται και την έκθεση Λάιον που ήταν ρήξη και έλευθη και νομίζω ότι πολλά από συμμερίζονται όλοι τις ε, απόψεις σου γιατί τώρα είσαι άλλη θέση αλλά όφυλα να τα πω αυτά. Περνάμε τώρα στη σε πολλά σημεία συμφωνούμε και θεωρώ ότι έχει νόημα η έκθεση πρωτοβουλίας μας να προηγηθεί της ίσως και το Μάιο να έχουμε την ε, τελική έγκριση στην Ολομέλεια για να προλάβουμε να το επιδώσουμε εγκαίρως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όρφος των πολιτικών και φυσικά θα πρέπει να εντρυφήσουμε στα θέματα της βιωσιμότητας και των κλιματικών αλλαγών αλλά καλό θα ήταν να συμπεριλάβει γιατί συνήθως ε, μιλούμε για την άμυνα και τις ενισχύσεις, αλλά ελάχιστα μιλούμε για τις αγορές που είναι τελικά. Αγαπητέ Άλμπερτ Όρφμαν, σε ευχαριστώ πολύ για τις βασικές κατευθύνσει ε, που περιγράφει η εκθεσή του. Είναι μια από στεναρό προπολογισμό για τη γεωργία. Σε αυτό πρέπει να κάνουμε περισσότερη προσπάθεια και βεβαίω είναι πολύ σημαντικό για μένα να μην λησμονούμε ότι έχουμε κοινή αγορά και μια κοινή πολιτική οπωσδήποτε χρειαζόμαστε εξ αυτού του λόγου. Βεβαίως δεν ε, μπορούμε να εγκαταλείψουμε το στόχο της ε, προμήθειας του Γεωργού και την διαφύλαξη της υπαίθρου των περιφερειών και της παραμονής των πολιτών σε αυτές και βέβαια το κλίμα, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Νομίζω ότι μπορούμε να αναπτύξουμε και περαιτέρω τομείς, ε, επί παραδείγματι το ζήτημα της πληρωμής από το πρώτο εκτάριο. Φορά τους νεαρούς γεωργούς μπορούμε να εξασφαλίσουμε κάποιες βελτιώσεις. Η κοινή γεωργική πολιτική δεν είναι ε, στα τελευταία της τα Ταλίστια. Πιστεύω ότι έχουμε τις δυνατότητες μέσα από την επικουρικότητα και με τις δυνατότητες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε τη δυνατότητα να τα καταφέρουμε. Είναι ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιήσουμε για να προσφέρουμε στις περιφέρειες ευελιξία. Πλην όμως για μένα και ως Γερμανίδα αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε αν χρειαζόμαστε τις εξαρτημένες, ε, συνδεδεμένες πληρωμές ε, και αντίστοιχα ζητήματα. Ε, ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την πρόταση και περιμένουμε δημονία την περαιτέρω συζήτηση. Καλούμαστε σήμερα ως Κοινοβούλιο να τοποθετηθούμε με μια πρώτη ιδέα, με μια πρώτη πρόταση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ βεβαίως θα πρέπει αυτό το οποίο θα προσδιορίσουμε να είναι κάτι το ορθό, να μην στρεβλώνει την κατάσταση, να μην είναι λάθος θεσμικό. Ιδιαίτερα για τον προπολογισμό, επιτρέψτε μου κάποια σχόλια, διότι ο Επίτροπο Έττιγκερ πρόσφατα μα μίλησε για περικοπέ στη Γεωργία, ειδικά 10 δισεκατομμυρίων. Αντί να μιλούμε για περικοπέ, πιστεύω θα ήταν πολύ καλύτερο να μιλούμε για εξοικονόμηση πόρων. Και άρα εκεί θα χρειαστεί μια προσεκτική ανάλυση του που πηγαίνουν τα ποσά, ώστε να περιοριστούν οι περιτές ε, δαπάνες, η διασπάθηση των κονδυλίων και να εξασφαλιστεί η εξοικονόμηση των πόρων και ταυτόχρονα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια σύγκληση ε, πραγματική των πληρωμών, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Είναι πολύ μεγάλες οι αποκλήσεις στον κοινωνικό ιστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι μια απόλυτη σύγκληση θα ήταν οπωσδήποτε άνηση και μάλιστα εις βάρος των γεωργών στα κράτη εκείνα όπου είναι πιο υψηλό το κόστος ζωής. Είναι απαραίτητο βεβαίως να διαφυλαχθούν οι δεσμοί μεταξύ της διτήρησης των πληρωμών και των δικτών ε, του μέσου κατακεφαλήν εισοδήματος, ώστε να μην καταλήξουμε σε συστήματα αθέμητου ανταγωνισμού. Βεβαίως πρέπει να κοιτάξουμε τις επιχειρήσεις που έχουν, ε, που έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες στις αγορές, περισσότερες δυσκολίες, μας μιλάει η πρόταση για την ε, βιομηχανοποίηση της παραγωγής που θεωρώ επικίνδυνη. Άρα οι πληρωμές θα πρέπει να ε, κυμαίνονται έτσι και να κλιμακώνονται έτσι ώστε να επιτρέπουν κίνητρα για κερδοσκοπία και σε, στην αγορά της γης των γεωργικών γεών. Πρέπει να βοηθήσουμε να συνδεθεί ο κόσμος της γεωργίας και στον ψηφιακό κόσμο, γιατί μπορεί πολύ ε, συχνά να φαίνεται πως ανήκει στο παρελθόν ε, ο κόσμος της γεωργίας, ότι είναι κολλημένος κάποιους αιώνες πριν, ενώ μπορούμε να αποδείξουμε ότι μπορεί να συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Χάρη στις, μεγάλες τεχνολογίες, νέες τεχνολογίες και τις μεγάλες περιόδους, μπορούμε να, να εξασφαλίσουμε ένα τομέα πολύ πιο αποτελεσματικό, παραγωγικό, σύγχρονο, αλλά και ικανό να προσελκύσει τη νέα γενναία Χαίρομαι ιδιαίτερω λοιπόν και ευχαριστώ τον εισηγητή για το έργο του και είμαι βέβαιος ότι ακόμη και με τις στενές προθεσμίες που μας έχετε ορίσει θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια πολύ καλή έκθεση. Μάλιστα, ακούσαμε τους και εισηγητές και τώρα περνάμε στους λοιπούς ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Τόρφμαν. την εισαγωγή του και της... Ε, την ε, χειρότερη περίπτωση θα πρέπει να δούμε αν θέλουμε επανεθνικοποίηση της ε, της γεωργικής πολιτικής, όχι, όχι τις ότι ας πούμε αφορούν στους έλεγχους, αλλά στην τελευταία μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής πολλές φορές είδαμε ότι καταλήγουμε σε πολύ μεγάλη γιατί κάποιοι λένε ότι α, γίνονται μόνο επενδύσεις για την γεωργία και άλλοι λένε ότι όχι γίνονται μόνο α, α, περιβαλλοντικές επενδύσεις. Σε κάποιους τομείς πραγματικά κατέληξαμε σε τέτοιες καταστάσεις, οπότε ας είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ναι, για το θέμα της επαναθνικοποίησης και εγώ να μιλήσω, ο κύριος Χόισλινγκ. Η Κομισιόν νομίζω θέλει να στείλει την ευθύνη σε άλλον. Δεν ε, καταφέρνουμε εμεί το στόχο, α να αφήσουμε στα κράτη-μέλη να τον επιτύχουν. Ε, νομίζω ότι ούτε ε, εγγυημένο εισόδημα καταφέραμε να πετύχουμε στους, για τους γεωργούς, ούτε οι αποδόσεις βελτιώθηκαν, τίποτα δεν καταφέραμε τελικώς. Αφού δεν τα πολύ μόνο εμεί, αφήνουν τα κράτη-μέλη μόνα του να καταφέρουν ό,τι μπορούν. Ε, για εμά, και τη Γερμανία θα είναι πολύ ε, μεγάλο το εγχείρημα αυτό αν θέλουμε από με 16 κρατήδια να βρούμε κοινό τόπο. Θα είναι πραγματικά πολύ επαχθής αυτή η διαδικασία. Οπότε εμείς πρέπει να αναλάβουμε την α, ε, ευθύνη και την Κομισιόν πρέπει να θέσει το πλαίσιο. Η ευθύνη πρέπει να είναι εδώ, στις Βρυξέλλες. Και επίσης να πω σαφώς, αν δούμε ποια είναι τα δύνατα σημεία αυτής της ε, προγραμματικής περίοδου, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να ισχύει πάντα η ίδια αρχή για την, ε, ναι, για την προστασία, των, ε, ε, για την ενίσχυση των προστατευόμενων αγορές. Το είδαμε, είδαμε τι γίνεται για, την, για τη ζάχαρη, είδαμε τι έγινε με το γάλα. Καταργούνται οι ε, κοινές οργανώσεις αγοράς, καταστρέφεται ο κλάδος. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν ε, κανόνες τους οποίους να μην μπορούμε να υπερβούμε για να πετύχουμε το στόχο μας. Ευχαριστώ. Ένα σύντομο σχόλιο. Μιλούμε για την γεωργία στην Ευρώπη. Και βεβαίως μιλούμε και για τα διάφορα μέσα που έχουμε στην, ε, διά, στη διάθεσή μας. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ξεχωριστή διαφορε, ε, γεωργική πολιτική για τις διάφορες περιοχές που υπάρχουν. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά βεβαίως ναι πρέπει να επιφέρουμε και μια αλφα ευελιξία στο πρόγραμμα. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ευχαριστώ. Πολύ σημαντική η συζήτηση αυτή. Θυμάμαι την ε, προηγούμενη φορά που, έκανα, που γινόταν αυτή η συζήτηση, ήμουν στο σπίτι μου και ε, έλεγα «Μα δεν νομίζω ότι έχουμε ε, καταλήξει τελικά στην αλήθεια, νομίζω ότι θέλω να εμπλακώ κι εγώ στη συζήτηση αυτή». Τώρα, υπάρχει μια αρχική δημόσια διαβούλευση η οποία λέει ότι 96% των πολιτών θεωρούν ότι η θέση του ε, παραγωγού στην ε, αλυσίδα διατροφής θα πρέπει να ε, ενισχυθεί. Και αυτό υπάρχει ένας πίνακας στις, στη σελίδα 14 που λέει ότι η Γεωργία βρίσκεται πολύ πίσω από άλλους τομείς. Δεδομένου λοιπόν αυτό, γιατί υπάρχει μόνο μία παράγραφο σε όλο αυτό το έγγραφο που αφορά ακριβώς αυτό το πρόβλημα γιατί αυτό είναι ο πυρήνα. Αυτό είναι η ουσία. Ανεξάρτητα από την υποστήριξη που θα δώσει κανεί. Τελικά καταλήγουμε να ε, ε, επιδοτούμε πολυεθνικέ. και ηλικιωμένου που δεν ανακατεύονται τόσο πολύ πια με την γεωργία. Υπάρχουν πολλά λοιπόν που πρέπει να συζητήσουμε, νέε τεχνολογίε, επενδύσει, νέο ρόλο για του γεωργού. Αλλά αν δεν υπάρχει εισόδημα για του ε, ε γεωργού τελικά, καμία διαφορά δεν θα είναι επιτυχία. Οπότε κάντε κάτι για το εισόδημα των ε, γεωργών. Είναι σαφές και είναι σημαντικό. Αλλά αν αυτό το σημαντικό θέμα το καλύπτουμε με μία παράγραφο... Βάζοντα ε, βάζοντας ε, λεφτά στην τσέπη κάποιου δεν κλείνουν τρύπε. Ο κύριος Κάρθη. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συμφωνήσω με το σχόλιο ότι αν αυτή η φάση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ ολοκληρωθεί χωρίς ε, ριζική επανισορρόπηση των ενισχύσεων της ΚΑΠ σε ό,τι αφορά την εξομοίωση και αποκατάσταση ισότητας μεταξύ των γεωργών, τότε θα έχουμε αποτύχει σε κάτι πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά το θέμα της επικουρικότητας και αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενδυναμώσει τα κράτη-μέλη. Εγώ συμφωνώ ότι όταν οι αποφάσεις ε, μπορούν να γίνουν σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καλύτερα να γίνονται εκεί. Αλλά υπάρχουν κάποια θέματα που θα μπορούν να γίνουν και σε επίπεδο κοινή γεωργική πολιτική. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις, όταν οι περιφέρειες και τα κράτη-μέλη ε, ε, λαμβάνουν ευθύνη για λήψη αποφάσεων, μερικέ φορέ θα κάνουν θάλασσα. Το, έχω, το γνωρίζω και εξ ίδιας Αλλά ε, το Ιρλανδικό Υπουργείο Γεωργίας πολλέ φορέ λέει στου παραπονούμενου γεωργούς ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συνήθως ε, υποβάλλεται το πρόβλημα σε εμά εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα λέει όχι, το πρόβλημα δεν ευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στην εθνική κυβέρνηση, στο Υπουργείο. Υπάρχει μια αμφισημία και στα διασταυρώμενα πυρά βρίσκονται εκλοβισμένοι γεωργοί. Αυτοί είναι οι χαμένοι. Επίσης να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε αυτή τη διαδικασία και όταν τα κράτη-μέλη έχουν συμπληρωματικές εξουσίες θα πρέπει να τις εκχωρούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογείται πρώτα και αυτό αντί να απαλείψει τη γραφειοκρατία, ίσως προσθέσει ένα ακόμη στρώμα γραφειοκρατίας. Το σημαντικό θα ήταν η Επιτροπή μας να καταθέσει τις σωστές τροπολογίες, ώστε να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Ο κύριος Σεράου Σάντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ντόρφαν. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι όπως είπα και προλαλήσαντες η Ευρωπαϊκή Γεωργία θα πρέπει να συνεχίσει να συμβάλλει στο, στη διατήρηση ενεργού πληθυσμού στην Ήπεθρο και να συμβάλλει στη αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας σε όλες τις περιφέρειες με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και με ενίσχυση της εδαφικής συνοχής. Οι μικρές εμβέλειες γεωργίας ε, και οι νέοι γεωργοί θα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο της πολιτικής για να πραγμα... καταφέρουμε να σταθεροποιήσουμε τον πληθυσμό της υπαίθρου και να καταπολεμήσουμε την απερίμωση. Σε ό,τι αφορά την πολιτική των αγορών, θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματικά μέσα για να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη αστάθεια των τιμών και της κρίσης και κυρίως να πατάξουμε τις αθέμετες εμπορικές πρακτικές που δημιουργούν στρέβλωση ανταγωνισμού. Ε, υπό την επιφύλαξη όλων όσων έχουν γίνει για το θέμα αυτό στον κανονισμό Omnibus. Τώρα, στο μοντέλο διαχείριση, αν αυτό προϋποθέτει μεγαλύτερη επικουρικότητα, θα πρέπει να συνδυαστεί με την μεγαλύτερη απλούστευση, τη λιγότερη περιπλοκότητα και την καλύτερη προβλεψιμότητα για τους γεωργούς και τις ε, εθνικές διοικήσεις, χωρίς να διακυβευτεί ο κοινό χαρακτήρας της κοινή γεωργικής πολιτικής. Γιατί αυτή τη στιγμή έχω πολλέ αμφιβολίες για τα θέματα αυτά, παρόλο που στόχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η απλούστευση. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω ω προ το νέο μοντέλο ε, παραγωγής. Πρώτον, πώς θα γίνει κοινό προγραμματισμός που θα συνδυάζει ταυτόχρονα ετήσια και πολυετή μέτρα. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει διαφορά στον ορισμό τι στη σφάλμα για τους ελέγχους και τις εποπτείες. Κάτι τέτοιο ε, ίσως ε, κάτι, ένα παρόμοιο πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί και σε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο που θα χαρακτηρίζεται με μεγαλύτερη επικουρικότητα, μεγαλύτερες διαφορές ερμηνείας δηλαδή. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι και από την ανακοίνωση της Επιτροπής ε, μπορεί κανείς να δώσει διαφορετικές ερμηνείες. Εσείς κύριε Ντόρφμαν, από ό,τι φαίνεται δώσετε την ερμηνεία ότι πρέπει να μείνουν τα πράγματα όπως έχουν. Ξέρω ένα βαθμό μπορώ να σας υποστηρίξω, αλλά εγώ διαβάζω διαφορετική ερμηνεία, ότι δηλαδή επιτέλους αλλάζουμε τη μπροστά. Λοιπόν, πάνω απ' όλα όμως υποστήριξη των μικρών και μεσαίων γεωργικών επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει ένα το επίπεδο, να υπάρχει μια σταδιακή με τη γεωργική πολιτική. Δεν, δεν ασχολούμαστε μόνο με του γεωργού, αλλά με την ύπεθρο γενικότερα και επίση θα ήταν σκόπιμο να κοιτάξουμε Έτσι λοιπόν, και αν προσανατολιστούμε στους στόχους, ε, το ότι πλέον δεν είναι μόνο γεωργική πολιτική. Έχουμε μπει στα βαθιά στην ανάλυση της ανακοίνωσης ε, του Επιτρόπου. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Νομίζω ότι ακριβώς σε χώρες με μεγάλη αποκέντρωση όπως η Ισπανία και η Γερμανία θα δημιουργήσει τεράστια περιπλοκή. Επίση, ό,τι αφορά τη μεταφορά των η χρηματοδότηση άλλων πολιτικών, όπως τη μετανάστευση από τη γεωρική πολιτική ή της αγροτικής ανάπτυξης από τη γεωρική πολιτική, είναι άδικη. Και ήδη να ξεχάσουμε και την ηλικιακή ανανέωση, αλλά και τη διαχείριση του κινδύνου. Ο κύριο Τάκουλα. Έχει κάποια θετικά στοιχεία και πρέπει από πλευρά μα να εξασφαλίσουμε τους όρους για άχθος για τον Ευρωπαίο παραγωγό και πρέπει να κοιτάξουμε και τον έλεγχο ή τόχους και αποτελέσματα. Είναι πολύ θετική, αλλά διαρωτώ με αυτά τα αποτελέσματα πώς θα ελέγχεται ότι έχουν επιτευχθεί και ότι διατηρούνται Και ασφαλώς πρέπει και οι στόχοι, οι κλιματικοί για τη γεωργία να είναι και αυτοί μέσα στο πρόγραμμα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρία Μακάρθη. Μαγκίνες. Ε, ευχαριστώ πολύ για την ε, τοποθέτηση του κύριου Ντόρφμαν. Οπωσδήποτε βέβαια το θέμα που μας απασχολεί είναι αν θα γυρίσουν όλες αυτές οι αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη και αν είναι τα κράτη-μέλη έτοιμα για να αναλάβουν αυτές τις αρμοδιότητες. Μπορεί κάποια να μπορούν, κάποια όχι. Τα διαθέσιμα ποσά. Ίσως θέλει ο εισηγητής μας να κάνει κάποιες διευκρινήσεις. Όταν μιλούμε για βελτίωση των στόχων, εννοούμε ασφαλώς ε, σύγκληση και ανώτατα όρια, οροφές. Ωστόσο αυτό θα σημαίνει ταυτόχρονα ότι οι πληρωμές του πυλώνα ένα θα αυξηθούν σε σχέση με των κρατών μελών θα διαμοιραστούν. Στην πράξη δεν ξέρω πώς θα υλοποιηθεί αυτό. Εγώ βεβαίως θα ήθελα από κάποια συστήματα να περάσουμε σε ε, ολοκληρωμένη ή ολιστική διαχείριση γεωργική. Υπάρχουν όμως και ενδεχομένως και άλλες λύσεις. Η, η διάσταση του πρασινίσματος από τελευταία κουγουπού και το έχω δηλώσει, αλλά ταυτόχρονα ίσως θα πρέπει να είμαστε ε, προσανατολισμένοι στη νέα αυτή ε, αναθεώρηση σε λύσεις που φέρνουν πραγματικά αποτελέσματα. Κυρία Κάντενμπαχ, προς ε, τελευταία να λέμε επικουρικότητα, ας γυρίσουν τα πάντα στα κράτη-μέλη, αλλά πρέπει να έχουμε και ένα είδους, ε, κατα... ενός είδους κατάλογο του τύπου αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη, γιατί ενδέχεται, αυτή την εντύπωση έχω εγώ τουλάχιστον, ότι κάποια κράτη-μέλη θεωρούν ότι θα κρατήσουν τα κονδύλια, αλλά θα τα διαχειρίζονται σε εθνικό επίπεδο και θα προσδιορίζουν μόνο τους θα τα κάνουν τα χρήματα αυτά. Να εξασφαλίζει ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα αξιοποιούνται κατά τρόπο αποτελεσματικό, κατά τρόπο εύστοχο για να μπορούμε και στο φορολογούμενο που λοιπόν πολλά ωραία συνθήματα ακούγονται ή τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως ακούγονται καλά. Ε, στη συνέχεια όμως πρέπει να ξέρουμε αν όντως επιφέραμε. Καλό αυτό, αλλά να μην ε, περιοριστούμε μόνο σε αυτό. Να δούμε το σύνολο τη πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που μου αρέσει στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι βελτιώσουν τη βιωσιμότητα σε επίπεδο αγροτική εκμετάλλευση. Να επικεντρωθούμε περισσότερο στι προσπάθειε, στι επενδύσει και στα αποτελέσματα που επέτυχαν οι Γεωργοί και να μην στη διαχείριση του κινδύνου και να βοηθήσουμε τους γεωργούς να παράσχουν αυτά τα πάντα. Ένα σύντομο σχόλιο. Η τρέχουσα ΚΑΠ είχαμε κάνει τις διάφορες επίσημες αλλά και άτυπες συμφωνίες για τη μεταρρύθμιση της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής. Ότι ας πούμε θα εξισορροπήσουμε το επίπεδο ε, άμεσων πληρωμών μεταξύ χωρών. Oui, merci, euh, Διαβάζω στην ανακοίνωση της Επιτροπής. Αισθάνομαι τον εξή φόβο και το ομολογώ. Σε οικονομική διασφάλιση του γεωργικού εισοδήματο, πάλι δεν προτείνεται τίποτα ούτε ουσιαστικό στον έγγραφο τη Επιτροπή. Και αυτό με ανησυχεί. Οι προοπτικέ με διαρκή μείωση του αριθμού των γεωργών και των γεωργικών εκτάσεων, μας οδηγούν, ε, φρονώ ότι πρέπει πολύ προσεκτικά να ε, μετρήσουμε τις επιλογές μας. Η κυρία Μαγκίνες μας ε, επεσήμανε πολύ σωστά της επιλογής μιας ασαφούς ομάδας στόχων, γιατί όσα πιο πολλά είναι τα επίπεδα της πολιτικής και θα, θα αυξήσουμε έτσι την περιπλοκότητα της όποιας μερωτικής πολιτικής και, την, και βέβαια θα είναι πολύ πιο δύσκολο να αξιολογήσουν, όπως είπε ο κύριος Βοητσικόσκι ή αλλιώς αν θέλουμε μια ουσιαστική, οπότε πρέπει αναλόγως να οργανώσουμε και τις εργασίες μας. Ευχαριστώ. Ακούσαμε όλους τους ομιλητές. Δεν έχουμε άλλον στο κατάλογο. Εγώ πιστεύω ότι η πρόταση μεταρρύθμισης της ΚΑΠ είναι περίπλοκη και απαιτεί μια διανοητική προσπάθεια και εκ μέρους των περιφερειών. Γιατί διατυπώνονται, κατάλο, διατυπώνονται στόχοι, αξίες, ε, ένας ολόκληρος κατάλογος με τέτοιους στόχους και αξίες. Και ε, θα πρέπει να έχουμε και τα αποτελέσματα όλων αυτών των προτάσεων. Να δώσουμε την ευκαιρία στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες να αποδείξουν ε, τι μπορούν να εφαρμόσουν. Και αυτό τα στρατηγικά σχέδια θα αξιολογηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είναι σημαντικό ε, όλα αυτά τα πράγματα να τα διεκπαιρεώσουμε πριν τις ευρωεκλογές. ώστε να έχουμε μεγάλη περίοδο συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών για την ε, ε, εκπόνηση των στρατηγικών σχεδίων. Γιατί αν αναβάλουμε τη σύντηση για αργότερα, θα μείνει πολύ, πολύ λιγότερος χρόνος για την ε, διενέργεια των στρατηγικών σχεδίων και την υλοποίηση αυτών των στόχων. Εγώ θεωρώ ότι είναι τεράστιο το επίπεδο των προκλήσεων. Είναι πραγματικά δυσθεώρητες αυτές οι προκλήσεις. Ε, έχουμε βέβαια μορφωμένους, καλλιεργημένους ε, γεωργούς, ε, διοίκηση επαρκώς τελεχωμένη. Είμαστε εξοικειωμένοι με όλα αυτά τα θέματα και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα για μια νέα προσέγγιση. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω ότι είναι δυνατή η μεταρρύθμιση. Είναι μεστή η πρόταση και καλό θα ήταν να έχουμε εμπιστοσύνη και να δείξουμε και λίγο θάρρος γιατί αν τα δούμε όλα αρνητικά, τα κράτη-μέλη θέλουν να είναι προετοίμαστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει τίποτα και η Γεωργία θα μας ξεγελάσει, τότε με τέτοια αρνητική προσέγγιση δεν θα πάμε πουθενά. Το λόγο έχει ο κύριος Μέγκελ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι θα τα είχα πει έτσι ωραία, όπως τα είπατε εσείς, Πρόεδρε. Πραγματικά ε, τονίσατε το πνεύμα της ε, ανακοίνωσης. Είναι μια προσφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και μια προσφορά προς το κοινό, προς τους πολίτες και οι ΚΑΠ συνολικά. Αυτή λοιπόν είναι η προσφορά η δική μας για να ξεκινήσει η συζήτηση και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Γιατί μιλούμε για την κοινή αγροτική πολιτική, η οποία ήδη είχε προτεθεί από την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή, ε, υιοθετήθηκε, μορφοποιήθηκε από τους νομοθέτες, από το Κοινοβούλιο δηλαδή και το μη ευθυνών μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού επίπεδου ή περιφερειακού επίπεδου. Η πρόταση δηλαδή είναι να αποσυρθούμε λίγο εμείς από το να ορίζουμε και να καθορίζουμε όλους αυτούς τους περίπλοκους κανόνες και στο παρελθόν και όπως το κάνουμε και τώρα και να δώσουμε την ευκαιρία στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες να βρούνε λύσεις πιο στοχευμένες για τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν που είναι και καλύτερα προσαρμοσμένες στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και βεβαίως που θα πληρούν πρόταση αναφέρθηκε η ανάπτυξη πέθρου που καλύπτει τους άλλους από το πρόγραμμα αλλά βλέποντας και τις άμεσες πληρωμές υπάρχουν περίπου 60 ή 70 διαφορετικές περιπτω... Ε, επιλογές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη. Ας πούμε την ε, συνδεδεμένη ενίσχυση. Έχουμε περίπου 200 προγράμματα. Ε, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι μονοδιάστατη αυτή η προσέγγιση. Είναι αρκετά ανομοιογενής με την καλή έννοια και περιλαμβάνει πολλές επιλογές. Αυτό προσπαθούμε λοιπόν να, να κάνουμε, να προσαρμόσουμε λίγο τους κανόνες της ανάγκης. τώρα, κάποια σχόλια για τα όσα ακούστηκαν και από μένα αντιμετωπίζει όλα αυτά τα ζητήματα και βεβαίως η Κομισιόν πολύ προσεκτικά παρακολουθεί το πώς μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα, πιο αυστηρά την αντιμετώπιση κινδύνου σε σχέση με το παρελθόν. Η θέση δηλαδή του γεωργού στον γεωργικό κλάδο ποια είναι και βεβαίως στα πλαίσια της ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της πολιτικής. Με έναν συνεκτικό τρόπο, συνεπή, αντί να έχουμε δύο πυλώνες, αλλά αυτό που θέλω να πω για να κλείσω είναι ότι βεβαίω έχετε απολύτω όλη τη στήριξή μα και όποια στιγμή χρειαστεί, χρειαστούν εξηγήσει από εμά, εμεί ευχαριστούμε να τι δώσουμε συμβολή στην όλη διαδικασία. Ο Επίτροπο βεβαίω παρακολουθεί πολύ στενά την, θα παρακολουθεί πολύ στενά τη συζήτηση που θα γίνει στην Επιτροπή σα και φυσικά είναι αποφασισμένο να το. Είναι σημαντικό να δούμε και την ουσία όλη αυτή τη μεταρρυθμιτική προσπάθεια και του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Γιατί ούτω ή άλλω και τα δύο αυτά